Uh, so, a very good afternoon, everybody, and a warm welcome to the European Parliament uh, for those come. Καλώς ορίσατε λοιπόν στην ακρόαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τελωνιακή εφαρμογή των ε, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα το οποίο επεξεργάζεται η Επιτροπή μας και είχαμε λοιπόν την αίσθηση ότι ήταν σημαντικό να ακούσουμε την άποψη και των εμπλεκομένων φορέων. Είμαι ιδιαίτερα ε, ευγνώμων στον κύριο Γιούργεν Κρόιτσμαν, ο οποίο είναι ο εισηγητή τη Επιτροπής που διοργάνωσε την ακρόαση αυτή. Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά μπροστά μα σήμερα το απόγευμα. Επιτρέψτε μου να αναφέρω κάποια ζητήματα για την διαδικασία ε, διοργάνωσης της ακροασής. Θα σας παρουσιάσει κάποιες λεπτομέρειες. Καταρχάς ο Γιούργεν Κρόιτσμαν για την πρόταση. Θα έχουμε τρία πάνελ. Το βλέπετε και στο πρόγραμμά σας. Τρεις ενότητες λοιπόν με εμπειρογνώμονες. Νομίζω ότι έχουν διαφορετικό χρόνο οι εμπειρογνώμονες στη διάθεσή τους. Α, όχι, 10 λεπτά maximum θα έχουν στη διάθεσή τους με χρονόμετρο. Φυσικά, αν δεν χρειαστείτε και τα 10 λεπτά, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Αλλά θα δώσω την ευκαιρία στους εμπειρογνώμονες να απαντήσουν στις ερωτήσεις που θα θέσουν οι υπόλοιποι. Τρεις ξεχωριστές, λοιπόν, ε, ε, ενότητες και μετά θα συνοψίσει ο εισηγητής. Ελπίζουμε οι άλλοι συνέδελφοι και κυρίως οι εισηγητές από τις χρηματοδοτούσες επιτροπές που ελπίζουμε να έρθουν θα πάρουν το λόγο αν το επιθυμούν. Αυτά λοιπόν ως προς την διαδικασία. Θα τελειώσουμε στις 6.30 το απόγευμα αλλά θα ήθελα καταρχάς να δώσω το λόγο στον Γιούργιν Κρόιτσμαν να σας πω ότι έχουμε διερμηνία στις ε, πιο πολλές γλώσσες. Επίσης να σας ε, ενημερώσω ότι η συνάντηση μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Ελπίζουμε να μας παρακολουθούν και όλοι οι δήμοι και οι κοινότητες που ενδιαφέρονται για τα θέματα αυτά. Δίνω το λόγο στον Γιούργεν Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάλκομ. Άκουσα ότι έχουν έρθει 50 ενδιαφερόμενοι σήμερα στην ακρόαση για την τελωνιακή εφαρμογή για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας. Χαίρομαι που είσαστε τόσο πολύ. Πρόκειται για μια οδηγία του 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία ορίζει πώς δραστηριοποιούνται τα τελωνία σε ό,τι αφορά ε, υποπτά προϊόντα για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι όροι είναι αρκετά τεχνικοί και δεν είναι πάντα αρκετά κατανοητοί. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό για μας ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ακούσουμε τους ειδικούς του κλάδου αυτού. Έχουμε λοιπόν σήμερα μια ευρεία γάμα εμπειρογνωμόνων από τον δημόσιο και τον δυτικό τομέα. Μαζί με τους υπάλληπους ε, εισηγητές αποφασίσαμε να γίνει μια διάκριση σε τρεις ενότητες. Την πρώτη ενότητα θα μας παρουσιαστεί πώς ε, τα εφιστάμενα τα ελληνιακά συστήματα θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Αυτό θα συμπεριλάμβανε τη διεύρυνση του τομέα εφαρμογή της υφιστάμενης οδηγία για νέες, να συμπεριληφθούν και νέε παραβιάσεις. Και εδώ τίθεται το ερώτημα κατά πόσον έχουν το δικαίωμα οι τρονιακές αρχές να δρουν παραπάνω. Επίσης, κατά πόσο οι αρχές αυτές μπορούν να αντιμετωπίσουν τις νέες διευρυμένες τους ε, ευθύνε με τα περιορισμένα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Επίσης, συγκεκριμένα ερωτήματα σε ό,τι αφορά τις μεταφορικές ε, εταιρείε και σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής συντοκτησίας. Επίσης, ποιος αναλαμβάνει την, ε, τον έλεγχο και το κόστος του ελέγχου. Αν αυτοί που καταστρέφουν τα προϊόντα θέλουν να αποζημιωθούν και διαπιστώνουν ότι η διεύθυνση παράδοσης ε, ήταν ψεύτικη και άρα δεν μπορούν να αποζημιωθούν. Να Επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσον δεν θα έπρεπε να επιτραπεί σε αυτούς που ζητούν αποζημίωση να προβαίνουν σε μεταφορές σε άλλα κρατημέλη για να γλιτώνουν κόστος. Χρειάζεται όμως και η έγκριση των τελωνιακών αρχών. Κατά πόσον δηλαδή ένα προϊόν το οποίο κατασχέται στο Λουξεμβούργο πρέπει να καταστρέφεται στο Λουξεμβούργο ή κατά πόσον θα πρέπει να μεταφέρεται σε άλλες ε, χώρες. Είναι ιδιαίτερη ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταστροφή των προϊόντων αυτών σε περίπτωση που υπάρχει διαπιστωμένη παραβίαση των ε, δικαιωμάτων πραγματική ιδιοκτησία. Δεύτερη ενότητα για τις επιδράσεις ε, στον καταναλωτή για τις ε, αποσκευές οι οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής. Υπό ποιους όρους όμως μπορούμε να μιλήσουμε για μη εταιρική χρήση. Αν κάποιος φέρει ένα ρόλεξ μαϊμού από τις διακοπές, είναι αποδεκτό εάν πρόκειται για ένα ρολόι. Ένα άλλο θέμα ε, που θα πρέπει να συζητηθεί είναι η ειδική διαδικασία για την ε, καταστροφή μικρών αποστολών. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει τραυματισμός του επιβάτη, του καταναλωτή, όταν ε, προβαίνουμε σε καταστροφή ενός ε, προϊόντος. Και δεν θα προκληθεί ζημιά στον καταναλωτή σε περίπτωση καταστροφής ενό τέτοιου προϊόντος. Πώς μπορούμε να ενημερώσουμε καλύτερα του καταναλωτές σε ό,τι αφορά τέτοια προϊόντα και επιπλέον δεν ορίζονται στο κείμενο της οδηγίας οι μικρές τέτοιες αποστολές, τα μικρά εμπορεύματα. Η Κομισιόν μας έχει δώσει 13 ορισμούς. Έχουμε ρωτήσει όλους τους ενδιαφερούμενους φορείς να μας βοηθήσουν και να μας πούν τι πιστεύουν. εκπροσωπούνται μόνο οι τελεμιακέ αρχέ και οι επιχειρήσει. Παρόλο που είχαμε καλέσει και ενώσει προστασία καταναλωτή. Δεν ξέρω γιατί δεν ήρθαν όμω, γιατί δεν ανταποκρίθηκαν, γιατί θα ήταν σημαντικό να ξέρουμε και την απόψη των καταναλωτών. Στην τρίτη ενότητα κοιτάμε τα εμπορεύματα, τα προϊόντα σε διαμετακόμιση σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάποιες περιπτώσεις τα τελωνία προέβησαν σε κατάσχεση προϊόντων τα οποία αποθηκεύονταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν προορίζονταν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ θα έχουμε υπόψη γενώσιμα φάρμακα προς, ε, που στέλνονται προς Ινδία και το καθεξής. ή τα οποία παράγονται στη Βραζιλία. Μια μικρή ερώτηση κατέθεσα και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ποιος ήταν ο λόγος εξαίρεσης από την οδηγία των προϊόντων αυτών. Η απάντηση ήταν ότι υπάρχει δυνατότητα να προβούν τα τελωνία σε κατάσταση. Άρα, το ερώτημα που ανακύπτει είναι, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα αυτή, μήπως θα έπρεπε να το διευκρινίσει η οδηγία. Μήπως όμως είναι αρμόδια και η Επιτροπή Ίντα. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τι πιστεύει και η Επιτροπή για το θέμα αυτό, η Επιτροπή Ίντα. Γιατί είναι ιδιαίτερα ο κίνδυνο των διερχομένων γεννόσιμων φαρμάκων ιδιαίτερα και θα πρέπει να υπάρξει καλύτερο ορισμό. Ελπίζω σήμερα να έχουμε και να βρούμε τις απαντήσεις στα πιο πολλά από αυτά τα ερωτήματα. Θα ήθελα να ακούσω και τους συναρμόδιους συζητητές. Δεν ξέρω όμως αν έχουν καταφτάσει. Η κυρία Γκάλο είναι εδώ, μάλιστα, πολύ ωραία. Να δώσω το λόγο. Σας ευχαριστώ. Αυτά εισαγωγικά. Okay. okay. Uh, very much indeed. Uh, yes, can I just uh, welcome... Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να καλωσορίσω τους συζητητές μας από τις επιτροπές με τις οποίες ε, έχουμε στενή συνεργασία. Έχουμε την ε, κυρία Άντρες Περέα από την ε, Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και την κυρία Γκάλο, η οποία είναι αρμόδια από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, είναι μέλος και της δική μας Επιτροπής. Νομίζω ότι θα δώσω το λόγο στην κυρία Άντρες Παρέα πρώτα. Αν θέλετε να κάνετε κάποια εισαγωγικά σχόλια. Τέσσερα λεπτά σας δίνουμε, maximum. Gracias. Eh, bueno, gracias por haber sido invitada a este σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων για αυτό το εξαιρετικά σημαντικό θέμα με το οποίο ασχολείται και η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, μάλλον ε, είναι αρμόδια επί της ουσίας. Μιλάμε για διεθνές εμπόριο Οπότε θα πρέπει να δούμε τη σύνδεση ανάμεσα στις παγκόσμιες τάσεις και το τι συμβαίνει στις μεμονωμένες οικονομίες μας. 0,04% του ΑΕΠ αντιστοιχεί αυτό το είδος εμπορίου. ο καταναλωτής θα πρέπει να μπορεί να χαίρει ε, διαφόρων δικαιωμάτων, θα πρέπει να προστατεύεται από την πειρατεία και την ε, παραχάραξη ε, και ο ρόλος των τελωνίων είναι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο την Επιτροπή ΙΝΤΑ. Το τελωνίο έχει ως ρόλο τον έλεγχο των εισαγωγών-εξαγωγών στα σύνορα. Σε εκείνη τη στιγμή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πλαστά προϊόντα. Πρέπει να ενισχυθούν τα τελωνία λοιπόν προς όφελος ε, της βιομηχανίας και της ανταγωνιστικότητας για να προστατευτούν τα σήματα και οι ευρεσιτεχνίες. Στην ουσία πρέπει να προστατευθούν οι επενδύσεις, η έρευνα και η καινοτομία. Και σε κοινωνικό επίπεδο ενθαρρύνεται έτσι η επασχόληση. σημαντικό στοιχείο στη στρατηγική της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δικαίω. Θα ήθελα τώρα να θίξω τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε. Νομίζω πως ήδη υπόθηκε αυτό. Είναι το θέμα των προϊόντων που είναι σε διέλευση, δηλαδή σε transit. Δεν είναι καταγεγραμμένα και δεν αποτελούν τμήμα του στόκ της κάθε επιχείρησης. Και αυτή η έννοια της διέλευσης προσφέρει ένα παράθυρο για τα ε, παραποιημένα προϊόντα, γιατί μπορεί να μπερδευτεί κανείς και να χαθεί μέσα σε αυτό το λαβύρινθο των διατυπώσεων. Έτσι μπορούν να μπουν ε, στην κοινότητα πολλά ε, παραποιημένα προϊόντα και θα αφιερώσουμε ένα μέγα τμήμα αυτής της συνεδρίασης σε αυτή την πτυχή. Μιλάμε για αυτά τα θέματα στην αιτιολογική έκθεση, αλλά εγώ θα ήθελα να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Τα παραποιημένα προϊόντα που βρίσκονται σε τράνζιτ θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο του ίδιου του νομοθετικού κειμένου. Να υπάρχουν γραφεία ελέγχου, ελέγχου κατά της απάτης, δραστηριότητες επίσης για την, που ασχολούνται με τη δημόσια υγεία και τις στατιστικές. Το προσωπικό δε αυτών των τελωνιακών γραφείων θα έχει ε, τέτοιο προσωπικό που το οποίο να είναι κατάλληλα καταρτισμένο για να μπορεί να ενεργήσει αντιπροσωπεύοντας το κράτος. Είναι δύσκολο όμως αυτό να γίνει στην πράξη. Υπάρχουν εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια. Εγώ προέρχομαι από την Βαλένσια, στην Ισπανία, όπου έχουμε λιμάνι με τεράστιες εισαγωγές εξαγωγές. Ο αριθμός των container ε, είναι τεράστιος και οι τελωνιακοί δύσκολα μπορούν να εντοπίσουν τα ύποπτα εμπορευματοκιβώτια. Σας μίλησα μάλιστα και να σας μιλήσω μάλιστα και για, μάλλον έγινε λόγος για τα φάρμακα γενικευμένης ονομασίας τα οποία επίσης μπορεί να είναι σε transit, μπορεί κανείς να τα παράγει, να τα παραποιήσει. Ε, είναι ένα προϊόν το οποίο πρέπει να παρακολουθηθεί γιατί μπορεί να παραποιηθεί πολύ εύκολα. Και ήθελα να επιμείνω στη διεθνή συνεργασία. Γιατί χάρη σε αυτήν μπορούμε να καταπολεμήσουμε την πειρατεία και την παραποίηση. Και πρέπει να το αναφέρουμε αυτό. Και εδώ υπάρχουν οι παράλληλες εισαγωγές. Θα πρέπει να μιλήσουμε για τις παράλληλες εισαγωγές, που δεν, ε, θέμα που δεν φαίνεται σε αυτό το έγγραφο, αλλά θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία λύση για την παραποίηση και την παραχάραξη των προϊόντων ε, εισαγωγής-εξαγωγής. Σας ευχαριστούμε, προσθέσατε κάποιες λεπτομέρειες και έχουμε ειδικά θέματα αργότερα όσον αφορά τα αγαθά σε τράνζιτ, σε διέλευση. Και τέλος να καλωσορίσουμε και την κυρία Γκαλό, η οποία θα μας δώσει την εικόνα από την οπτική γωνία της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω πως αυτή η ακρόαση είναι εξαιρετικά χρήσιμη, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να ακούσουμε τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων, των επιχειρήσεων, των τελωνιακών αρχών για τον τελωνιακό κανονισμό κατά της παραπίσης και να διαρωτηθούμε για τεχνικά θέματα αλλά και για πολιτικά ευαίσθητα ζητήματα τα οποία θα αναφέρω στη σύντομη μου εισήγηση. Να διευκρινίσω ότι όσο με αφορά εγώ έχω διπλή ιδιότητα, γιατί όπως είπατε είμαι η εισηγήτρια για γνωμοδότηση στην Ζούρη, αλλά είμαι και σκιώδηση εισηγήτρια του ΕΛΚ στην ΙΜΚΟ. Πολύ σύντομα λοιπόν τρεις παρατηρήσεις. Καταρχήν για το πεδίο εφαρμογής. Όπως μόλις άκουσα τη συνάδελφό μου, ε, έχει προβληματίσει όσον αφορά τις παράλληλες εισαγωγές. Θα πρέπει να καλύπτονται από τον μελλοντικό κανονισμό. Πρόκειται για ε, μία διαφορά που προκύπτει από κάποια συμβατική σχέση ή πρόκειται για παραβίαση ενός δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας που απαιτεί την παρέμβαση των τελωνιακών αρχών. Η Κομισιόν μας προτείνει τη διατήρηση μάλλον δεύτερος προβληματισμός. Η Κομισιόν μας προτείνει να διατηρήσουμε την εξαίρεση των ε, μπορευμάτων που, που περιέχονται που, που μάλλον βρίσκονται μέσα στις προσωπικές αποσκευές των επιβατών. Μπορούμε να δεχτούμε ότι ένας τουρίστας ο οποίος ε, επιστρέφει από την Κίνα φέρνει τέσσερις τσάντες βουητών και αυτός να μην ελεγχθεί, ενώ αυτός ε, που θα του στείλουν ένα με το, μία τσάντα τέτοια με το ταχυδρομείο να ελεγχθεί αυστηρά από τον νόμο. Ξέρω πως αυτό το ερώτημα δεν είναι πολιτικό ορθό και ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να παραδεχτεί κανείς ε, τα προσωπικά, οι προσωπικές αποσκευές να μην ξεφεύγουν από αυτό το κανονισμό. Δεύτερον, όσον αφορά τα ε, φάρμακα γενικευμένης ονομασίας και εδώ είναι ένα πολιτικό ζήτημα εξαιρετικά λεπτό και λόγω της εμπορικής ε, διαφοράς ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ινδία και τη Βραζιλία. Στην νομοθετική, υπηρεσία έχουμε ένα, στην νομοθετική πρόταση έχουμε μια, ένα εκτιμώντα υπαριθμό 17 και σύμφωνα με την άποψη τη Κομισιόν είναι παρκέ αυτό για να ρυθμίζονται οι διαφορέ. Ελπίζω πω οι παρεμβαίνοντε ω προ αυτό θα μα δώσουν κάποιε διευκρινήσει. Προσθέτω ότι τα παραπημένα φάρμακα έχουν άμεση σχέση με τη δημόσια υγεία. Διαπιστώνω διαβάζοντας το πρόγραμμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα παραπημένα φάρμακα ότι όντως σε πάρα πολλές αφρικανικές χώρες ή χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής και μάλιστα στις χώρες που υπάρχει οικονομία μετα... μετάβασης, εκεί η αναλογία ε, παραπημένων φαρμάκων είναι η πιο υψηλή. Αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη από το νομοθετικό κείμενο. Τρίτη παρατήρηση με τη σειρά μου για τις μικρές, τα μικρά ταχυδρομικά δέματα. Όπως γνωρίζετε, το ταχυδρομική κίνηση, εκεί οι κατασχέσεις έχουν ε, πολλαπλασιαστεί κάθετα. Από τις 15.000 στάσανε στις 83.000 το 2009. 10, ε, με συγχωρείτε. Επ' αυτού η Γαλλία έχει φτιάξει μια ελαφριά διαδικασία για την αντιμετώπιση των μικρών ποσοτήτων ε, παραποιημένων προϊόντων στον τομέα των δεμάτων express και των ταχυδρομικών δεμάτων. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψη των ε, παρεμβαινόντων για την διαδικασία που προτείνει η Κομισιόν. Θα είναι αποτελεσματική για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και η προθεσμία 20 εργάσιμων ημερών που προβλέπεται αυτή τη στιγμή από το άρθρο 24 είναι σύμφωνη με τον απλό χαρακτήρα που θα πρέπει να έχει μια τέτοια διαδικασία. Αυτά κύριε Πρόεδρε, κάποιες ε, στοιχεία που νομίζω ότι είναι σημαντικά και που θα επιτρέψουν να τροφοδοτηθεί η συζήτηση την οποία θα ακούσαμε με μεγάλη προσοχή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ και τους δύο και βεβαίω ε, θα περιμένουμε τα σχόλιά σας. Τώρα προχωράμε στον, στην πρώτη συνεδρίασή μας για την εξασφάλιση του σωστού τελωνιακού ελέγχου. Όλοι έχετε αντίγραφα των βιογραφικών των ομιλητών, δεν θα σας μιλήσω για αυτούς. Λοιπόν, θα ακούσουμε πρώτα απ' όλα τον, τον Κριστόφ Ζίμερμαν. Τον καλωσορίζω ιδιαίτερα θερμά γιατί τον πρωτοσυνάντησα όταν δούλευε στην Κομισιόν για την τελωνία, στον τελωνιακό έλεγχο. Ασχολείται τότε με την κεραμική βιομηχανία. Τώρα είναι στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνίων και έχει πολύ σημαντική θέση. Μας έχει βοηθήσει πάντα και είναι ο ιδανικός άνθρωπος για να ξεκινήσει σαν ομιλητής σε αυτό το τις συνεδρίες. Κριστόφα, έχεις το λόγο. Δέκα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Πριν από 12 χρόνια, κύριε Πρόεδρε, ακριβώς ασχολούμαι με τα παραποιημένα κεραμικά, αλλά όχι μόνο. Πράγματι. Υπάρχει και παραποίηση όμως και πλαστά στην κεραμική. Σας ευχαριστώ που δίνετε το λόγο στον οργανισμό, το Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνίων 177 διοικήσει εκπροσωπούνται. Βεβαίω, εμεί γνωρίζουμε καλύτερα τα όσα συμβαίνουν στα διεθνή σύνορα. Στην εντολή του οργανισμού του τελωνίων δεν έχουμε τη δυνατότητα να κρίνουμε αν είναι αιτιολογημένη μια νομοθεσία ή όχι, ή μια πρόταση νομοθετική. Όμως θα ήθελα να επιμείνω για δύο τάσει οι οποίε αναδύονται εδώ και μερικά χρόνια, τρία-τέσσερα χρόνια μάλιστα. Έχουμε παραβιάσεις και μιλάω για παραποιημένα προϊόντα τα οποία θίγουν την υγεία. Λοιπόν, έχουμε παραβιάσεις της πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά έχουμε και επιπτώσεις της παραποίησης σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτό το λαθρεμπόριο θα έλεγα το ταχυδρομικό λόγω του, του διαδικτύου θα βρει τη λύση του. Έχουμε πάνω από τρία δις ταχυδρομικά δέματα που κινούνται κάθε χρόνο και κάτω από ένα εκατομμύριο τελωνιακού στον κόσμο. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι να παρεμποδιστεί αυτή η ροή, η λαθρέα ροή. Το πρόβλημα αυτής της πειρατείας των παραποιημένων προϊόντων είναι εξελικτικό. Δηλαδή, οι διαδρομές της απάτης αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε πολλά θέματα σε μεταφόρτωση, σε τράνζιτ, η έλευση δηλαδή, η αλλαγή εμπορευμάτων στην ελεύθερη ζώνη όπου δεν υπάρχει έλεγχο, έλεγχος, δηλαδή ακολουθούμε το κοντέινερ, τον αριθμό του, αλλά δεν έχει το ίδιο εμπόρευμα μέσα. Έχουμε εξελικτική λοιπόν τάση ακόμη ε, στη διακίνηση, αλλά και στα ίδια τα προϊόντα. Εκτός από τα προϊόντα πολυτελείας, έχουμε και άλλα θέματα. Σε τρεις μέρες ε, στην Αφρική βρήκαμε 43 εκατομμύρια παραποιημένα προϊόντα. 5.000 ήταν τσάντες πολυτελείας και 8 εκατομμύρια ήταν ε, φάρμακα. Λοιπόν, αυτό το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι όταν μιλάμε για παγκοσμιο, παγκοσμιοποίηση. Το ίδιο συμβαίνει και με την απάτη. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ευρώπη ή στον κόσμο δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει μόλις βγούμε από την Ευρώπη. Πάντα υπάρχει κίνδυνος επιστροφής μέσω του διαδικτύου, διότι σήμερα όσον αφορά την παραποίηση και όχι την πειρατεία, δεν έχουμε από του αντικειμένου Το παραποιημένο φάρμακο, το παραποιημένο τρόφιμο μεταφέρεται ταχυδρομικά. Το πρόβλημά μας δεν είναι το διαδίκτυο. Το πρόβλημά μας είναι η πολλαπλότητα, ο μεγάλος αριθμός των δεμάτων που φτάνουν τη νύχτα, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε ανάλυση κινδύνου τη νύχτα, διότι δυστυχώς ε, δεν έχουμε σύστημα προειδοποίησης τη μόνη τεχνική που έχουμε στο ταχύδρομείο είναι να, κοπ... να ανοίξουμε ένα δέμα και όταν έχουμε τρία δις δέματα είναι δύσκολο να κάνει κανείς μια σωστή ανάλυση. Πρόεδρε, επιτρέψτε μου επίσης να επιμείνω σε δύο-τρία θέματα. Έχω κάποιες φωτογραφίες για να σας δείξω. Εδώ έχουμε παραποίηση παπουτσιών που φτάνουν στην Ευρώπη, γιατί τα βρήκαμε στην Ιταλία. Είναι τοξικά παπούτσια. Είναι μια παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησία, αλλά για δέστε και τι γίνεται με την δημόσια υγεία. Κοιτάξτε πώ γίνονται τα πόδια όταν τα φορέσετε. Λοιπόν, εδώ έχουμε συστήματα ανείχνευση πυρκαγιά. Παραποιημένα Πώς το ανακαλύψαμε, ένα ξενοδοχείο στο Κουβέιτ και ολόκληρο, παρόλο που είχε αυτούς τους μηχανισμούς. Λοιπόν, μιλάμε πλέον για παραποίηση η οποία παραβιάζει την υγεία και την ασφάλεια του καταναλωτή. Εδώ έχουμε κρέμες που δεν υφίστανται. Με συγχωρείτε που βλέπετε τις μάρκες, αλλά είναι αρκετά εντυπωσιακό. Αριστερά, δεξιά σας δηλαδή κύριε Πρόεδρε, έχουμε μια πολύ γνωστή μάρκα κρέμας που σε αυτή την περίπτωση ε, είναι για την αύξηση των μειών ε, του στήθους. Τι να σας πω, βεβαίω η μάρκα αυτή ποτέ δεν παρασκευάζει τέτοιου τύπου κρέμες, αλλά βλέπετε, ε, αυτό μπορείτε να το βρείτε και στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης. Εδώ δεν σας δίνουμε τη μάρκα, αλλά ε, δέστε τι ανακαλύπτουμε παντού πώς γίνεται μια, ένα πολύ γνωστό ποτό, ε, αναψυκτικό μάλιστα, ευρεία κατανάλωση. Ορίστε πώς κατασκευάζεται. Λοιπόν, ε, χρειάζονται πρωτοβουλίες και από την Κομισιόν και από τα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε νομοθετικά με το φαινόμενο, στο φαινόμενο μάλλον. Ε, ο τελευταίος κανονισμός ήταν το 2003. Μέχρι το 2011 έχουν αλλάξει τα πάντα είναι εξελικτικά. Θα σας δώσω κάποιους αριθμούς. Συν 600% παραποίηση μεταξύ 2002 και 2008 για τα τρόφιμα, 127% για τα ανταλλακτικά, 19% αύξηση στις κατασχέσεις για τα φάρμακα. Ε, πρέπει να ξεχωρίζουμε τα πλαστά από τα παραποιημένα. 2009-2010, 110% αύξηση της παραποίησης τροφίμων και οι στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ταξιούτ επιβεβαιώνουν. 10.000 περιπτώσεις είχαμε το 2003 στα σύνορα. 79.000 το 2010, δηλαδή έχουμε 7 φορές παραπάνω διαδικασίες κατάσχεσης και τα λοιπά για παραποιημένα. Όλα αυτά οφείλονται και στο διαδίκτυο. Ξέρετε το 2008 έγινε μια σημαντική επιχείρηση σε 27 κράτη-μέλη, η Medifake. Αυτή η επιχείρηση είχε οδηγήσει σε 34 εκατομμύρια φάρμακα που ανοιχνεύτηκαν παραποιημένα. 34 εκατομμύρια παραποιημένα. Αυτό σημαίνει βέβαια παραχαραγμένα, αλλά μέσα σε δύο μήνες έγινε αυτό. Η διαπίστωση αυτή. Η επιχείρηση Παντζέα της Ιντερπόλ επιβεβαιώνει αυτό το φαινόμενο. Εν ώψη όλων αυτών λοιπόν θέλουμε να σας παροτρύνουμε και να σας ενθαρρύνουμε να ενισχύσετε την νομοθεσία να ανταποκρίνετε στην πραγματικότητα γιατί έχουμε μία πανδημία δεν μπορούμε να βάλουμε ένα τελωνιακό πίσω από κάθε κοντέινερ, πίσω από κάθε αεροπλάνο, πίσω από κάθε ταχυδρομικό δέμα. Αλλά μέσα στο σημερινό οικονομικό πλαίσιο έχουμε προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Έχουμε την ασφάλεια και την υγεία του καταναλωτή, αλλά έχουμε και την οικονομική πρόκληση, διότι το μερίδιο της αγοράς που καταλαμβάνουν τα παραποιημένα ε, έχει επιπτώσεις για τις χώρες μας. Τέλος, πρέπει να βρούμε μια οριστική, δραστική λύση για το διαδίκτυο και τα ταχυδρομικά δέματα. Καταλήγοντας, σας δείχνω μια άλλη εικόνα, παραποιημένα τηλεφώνα, κινητά, τα οποία εκρήγνεται. Είναι αληθινές φωτογραφίες αυτές, κύριε Πρόεδρε. 500 τόνοι παραποιημένο αντομοκτώνα. Πράγματα τα οποία δεν βλέπουμε, αλλά τα οποία εισπνέουμε. Αυτά τα βρήκαμε στα σύνορα βέβαια και θα τελειώσουμε αυτές τις εικόνες. Η παραποίηση σκοτώνει. Λοιπόν, δεν προσπαθούμε τώρα να προκαλέσουμε γενικό συναγερμό, αλλά κοιτάξτε τι βρίσκουμε σε ένα φαρμακείο. Εμβόλιο παιδιατρικό. Βλέπετε τώρα ότι πάνω στη βελόνα έχουμε κομμάτια από αίμα, ίχνη από αίμα μάλλον και από δέρμα και αυτό πωλείται για να εμβολιαστούν παιδιά και έχει μέσα το περιεχόμενο είναι απλά νερό. Λοιπόν, αυτές τις εικόνες μας τις δώσανε από μία ένωση, αλλά όταν μιλάμε για την παγκοσμίωση, πρέπει να σας πω ότι βρήκαμε μία οδοντόκρεμα σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ στην Αμερική. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα στα δόντια χρησιμοποιώντας αυτή την οδοντόκρεμα περιλαμβάνει μια καρκινογενή ουσία και αυτό το παιδί Απλώς έπαθε αυτό το καρκίνο που βλέπετε στο πρόσωπό του από αυτή την οδοντόκρεμα. Λοιπόν, είναι φοβερά όλα αυτά. Τώρα, το διαδίκτυο, μια υπόθεση δύο-τριών ετών. Pharmacy Online, το αποτέλεσμα αυτών που βρήκαμε. Ένα προϊόν έφυγε από την Κίνα, 450 κιλά, ε, αντικαρκυνικού φαρμάκου για την οστεοπόρωση λοιπά. Ξεκίνησα από την Κίνα, πήγε στο Χονγκ Κονγκ, πέρασε από το Ντουμπάι. Από το Ντουμπάι συνέχισε τη Μεγάλη Βρετανία και τελικός προορισμός οι Μπαχάμες. Το ανείχνευσαν στη Μεγάλη Βρετανία. Κατευθυνόταν για το εμπόριο στο διαδίκτυο. Τα 450 κιλά λοιπόν αυτά σταμάτησαν στη Μεγάλη Βρετανία είχαν προορισμό τις Μπαχάνες. Μπαχάμες. Στόχος ήταν η Αμερικανική αγορά. Ήταν αδύνατον να, ε, αυτοί οι απαταιώνες να στείλουν το εμπόρευμα στις Ηνωμένε Πολιτείε. Γι' αυτό έφτιαξαν μια φάρμαση online, ένα φαρμακείο online στον Καναδά, Μπαχάμες Καναδάς, Μεγάλη Βρετανία και επιστροφή. Αυτό είναι το πρόβλημα της ε, παγκοσμιοποίησης και το μετωπίζουμε όλοι γιατί πρόκειται για μικρούς φακέλους που φτάνουν στον πελάτη. Αυτή τη μαρτυρία είχα να σας δώσω, χωρίς να προκρίνω την πρωτοβουλία σας. Θέλω απλώς να ευαισθητοποιήσω το κοινό για το πόσο επικίνδυνα είναι όλα αυτά στα σύνορά μας. Ευχαριστώ. Well, thank you σας ευχαριστώ κύριε Τσίμερμαν και θα πρέπει να πω ότι ήταν τόσο εντυπωσιακά αυτά που μας λέγατε που δεν σας δίκοψα καν όταν ξεπεράσατε το χρόνο σας. Δεν πρόκειται αυτό να γίνει και για τους άλλους ομιλητές απαραίτητα, αλλά ε, νομίζω ότι ήταν πολύ προφανές το γιατί χρειαζόμαστε ε, αυτή την νομοθεσία. Θα περάσουμε τώρα στον κύριο Τζερεμί Νιούμαν, ο οποίος είναι ε, δικηγόρος σε θέματα της Επιτροπής κατά της παραχάραξης, κατά της παραποίησης. Σας δίνω το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, και καταρχά για την ευθύνη, την ευκαιρία να μιλήσω σήμερα το απόγευμα και ευχαριστώ, Κρίστοφ, που μας παρουσίασε το θέμα αυτό με τόσο έντονα παραδείγματα. Εγώ θα σας μιλήσω από την ε, Διεθνή Οργάνωση με 600 μέλη εκ των οποίων τα πιο πολλά είναι μέτρα στην Ευρώπη, τη Ρωσία και την CIS. Τρεις βασικές αρμοδιότητες έχουμε. Καταρχάς ενημέρωση και ε, δημοσίευση, ε, εκπαιδευτικά εκδηλωτικές εκδηλώσεις και ανάπτυξη πολιτικής. Ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι η προώθηση των ε, επωνυμιών και η προστασία των επωνυμιών για να μπορούμε να διασφαλίσουμε στον ε, καταναλωτή ότι ε, λαμβάνει αυτό για το οποίο πληρώνει. Η καταπολέμηση της παραποίησης αποτελεί ένα βασικό στόχο της ΙΝΤΑ. Ε, Μιλάμε για θέματα επωνυμίας λοιπόν και καταπολέμησης της παραποίησης. Ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο ζητά και χρειάζεται μία παγκόσμια λύση. Θα πρέπει να γίνει μία σωστή ανάλυση, να δούμε κατά πόσον το σχέδιο κανονισμού θα μας ε, οδηγήσει σε αποτελεσματική τηλεμιακή εφαρμογή και ιδιαίτερα κατά πόσο η πρόταση θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλει αποτελεσματικά στις προσπάθειες καταπολέμησης της παραποίησης. Γενικά, επικρατούμε τα βήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του κανονισμού και έχουμε προετοιμάσει λεπτομερή σχόλια. Στα 10 λεπτά θα εστιαστώ σε τέσσερις ε, διαφάνειες. Καταρχάς, ε, σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή και τους πόρους, ο υφιστάμενος ε, κανονισμών περιορίζεται στις παραποιήσεις, αλλά όχι σε άλλες μορφές παραβίασης και παράλληλες εισαγωγές. Γίνεται πρόταση να συμπεριληφθεί πιο ευρύ φάσμα παραποιήσεων και να αφαιρεθεί η εξαίρεση των παράλληλων εισαγωγών. Γιατί φυσικά υπάρχει και ανάμειξη των πρωτότυπων με τα παραποιημένα προϊόντα. Και αυτό θα έχει αντίκτυπο σε αυτούς που παράγουν τα παραποιημένα προϊόντα. Να σας πω ότι η Ένωσή μας ανησυχεί γιατί μπορεί να αποδυναμωθούν ενδεχομένω οι προσπάθειές μας αν δεν υπάρχουν επιπλέον πόροι. Να σας μιλήσω για την διαμετακόμιση επίσης, το οποίο θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε στα πλαίσια του τομέα εφαρμογή τη κανονισμού, επειδή είναι σαφέ ότι δεν πρόκειται να αλλάξει το επίπεδο, το κείμενο για τις παραβιάσεις. Υποστηρίζουμε την ε, κατάσχεση των παραποιημένων προϊόντων οποτεδήποτε και αν υπάρχει ευκαιρία και οποιοδήποτε και αν είναι ο προορισμός τους. Απλοποιημένη διαδικασία. Ε, καλωσορίζουμε την ε, υποχρεωτική απλοποίηση της νομοθεσίας. Να λάβουμε υπόψη τρία ζητήματα. Καταρχάς ότι οι υποεύθυνη παραποίηση, σπάνια είναι σε πρόθυμη να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους. Τα τελωνία, λοιπόν, όπου δεν λαμβάνουν απάντηση, θα πρέπει να θεωρούν ότι ο παραγωγός συμφωνεί για την ε, καταστροφή των προϊόντων. Κατά δεύτερον, προτείνουμε ο δικαιούχος να μπορεί να καταβάλει την αίτηση για καταστροφή των προϊόντων κατά τρίτον η ΙΝΤΑ θέλει να τονίσει ότι η απλοποιημένη αυτή διαδικασία μπορεί να είναι, μπορεί γρήγορη και ακριβή. Αλλά αν θέλουμε να είναι αποτελεσματική η νομοθεσία, θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο τα διοικητικά, οι διοικητικές κυρώσεις ε, έχουν αποτέλεσμα. Να σας ενημερώσουμε ότι οι δικαιούχοι κατανοούν τη σημασία της δημιουργίας μιας σχέσης με τα τελωνία, η οποία θα πρέπει να βασίζεται σε αμοιβαία κατανόηση και ανταλλαγή πληροφοριών. Η ίντα ανησυχεί ότι η πρόταση που έχει ως σκόπο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενδεχομένως να φέτει υπερβολικό βάρος στους δικαιούχους γιατί απαιτείται να παρέχουν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία στα τελωνία. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευρύ, γιατί κάθε λεπτομέρεια θα μπορούσε να θεωρηθεί σχετική. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε οι υποχρεώσει των δικαιούχων να εξισορροπούνται και να την υπόψη οι περιορισμένοι πόροι του. Επίση, ε, η ΙΝΤΑ θεωρεί ότι θα πρέπει να χορηγούνται και πληροφορίες στους δικαιούχους και να διέπονται από μία απαρέκλητη υποχρέωση να τις αντιμετωπίσουν με απόρτο τρόπο. Επίσης, θα πρέπει να καταπολεμάται και να αποτρέπεται η συμπεριφορά εμπορίας σε παραποιημένα προϊόντα. Το άρθρο 18 διευκρινίζει δεν διευκρινίζει να χορηγούνται πληροφορίε σε υπηρεσίε άλλων κρατών μελών, όπω η Τελωνία ή σε μέρη τα οποία είναι υπεύθυνα για την παραβίαση. Θεωρούμε ότι όταν διαπιστωθεί παραποίηση, μέσω της απλοποιημένης διαδικασίας, για παράδειγμα, η προστασία πληροφοριών σχετικά με τους εμπλεκομένους φορείς θα πρέπει να καταπίπτει. Τέλος, να στραφώ σε θέματα ευθύνης και κόστους. Η έλλειψη ε, σαφήνειας δίνει ευκαιρίες σε όσους ε, κάνουν κατασχέσεις ε, τέτοιων δεμάτων να προβαίνουν σε υπερβολικές κατασχέσεις. Εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη το άρθρο 27 το οποίο διευκρινίζει ότι δεν ε, ε, αναιρείται έτσι το δικαίωμα του δικαιούχου να ζητάει αποζημίωση, γιατί οι κυβερνήσεις χάνουν έσοδα, διακυβεύεται η υγεία των καταναλωτών και οι, εργατικές, οι συνθήκες εργασίας των ε, εργαζομένων. Γι' αυτό λοιπόν ο, φόρτος αυτός, το φορτίο αυτό θα πρέπει να κατανέμεται σωστά από αυτούς που εποφελούνται έμεσα ή άμεσα από την μεταφορά και την αποθήκευση των ε, εμπορευμάτων αυτών. Η Ένωσή μα θεωρεί ότι θα πρέπει να επιβληθούν σοβαρέ κυρώσει για οποιονδήποτε δεν αποφασίσει να εκκινήσει διαδικασία για να καθοριστεί κατά πόσον υπήρξε παραβίαση. Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να τιμωρούνται για να μην, όταν δεν επιλέγουν να καταγγείλουν μια περίπτωση λόγω του υψηλού κόστου, για παράδειγμα όπως του δικαστικού, των ε, δικαστικών εξοδών. Θα ήθελα να πω ότι τα υπόλοιπα βασικά ζητήματα θα μπορέσουν να εξεταστούν στην παρούσα φάση και φυσικά είμαστε επιτεθειμένοι να σας παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες σε περίπτωση που το επιθυμείτε και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μας καλέσατε σήμερα. Uh, Σας ευχαριστώ για την πολύ σαφή αυτή παρουσίαση και θα ήθελα να πω ότι έχετε τις διαφάνειες στο φάκελό σας. Και τώρα να περάσουμε λοιπόν στο Μαρκ Φραντεπέχ, ο οποίος είναι σύμβουλος για θέματα πολιτικής, τελωνικής πολιτικής μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μεταφορά και τις τελωνιακές υπηρεσίες για να μας μιλήσει για την οπτική γωνία ενός σημαντικού φορέα στο διεθνές προσκήνιο. Έχετε το λόγο. Thank you, for... Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να κάνουμε εδώ τις παρατηρήσεις μας. Cat, uh, is... Αντιπροσωπεύω την Κλέκατ που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ευρωπαϊκό, Ευρωπαίων Αντιπροσώπων για τις μεταφορές και τα τελωνία. Πρόκειται για μια διεθνή οργάνωση, μη κερδοσκοπική, που είναι καταγεγραμμένη στο Μητρό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπροσώπων συμφερόντων και όπως σας είπα αντιπροσωπεύουμε τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που προσφέρουν μεταφορικές υπηρεσίες, υλικοτεχνική υποδομή εντός και εκτός Ευρώπης. Θα πρέπει να σημειώσετε να σημειωθεί μάλλον τι είναι ένας ε, προωθητής φορτίων καθώς ε, παρέχουν ε, τις υπηρεσίες τους οι φορείς αυτοί ενεργούν εξ ονόματος των πελατών τους ποτέ δεν παίρνουν αποφάσεις σε σχέση με την εμπορική συναλλαγή ανάμεσα στον πολιτή και τον αγοραστή λαμβάνουν οδηγίες ή από τον έναν ή από τους δυο και από τους δυο, τις οποίες εκτελούν έτσι ώστε να καταστεί δυνατή εμπορική συναλλαγή χωρίς να υποκαθιστούν ε, τα συμβαλόμενα μέρη ε, μιας σύμβασης. Το Μάιο του 2010 η Κλέκα είχε τη δυνατότητα να συμβάλλει στη δημόσια διαβούλευση της Κομισιόν για την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και η παρέμβασή μας ε, εστιάστηκε απόλυτα στις ευθύνες των μερών που είναι οι ενδιαφερόμενοι στην ε, αλυσίδα παροχής προμηθειών, χωρίς όμως να εμπλέκονται στην εμπορική συναλλαγή. Ιδιαίτερα εξετάσαμε ποιο θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τα δικαιώματα πνευματική διοκτησία και το σχετικό κόστο, δηλαδή ποιο θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση και την καταστροφή αγαθών που παραβιάζουν τα δικαιώματα ε, πνευματική ιδιοκτησία. Καθώ και σε ποιο. Ε, το όνομα και προς το συμφέρον ποιου γίνεται η αποθήκευση ή και η καταστροφή αυτών των αγαθών. Σήμερα διαπιστάνουμε με ικανοποίηση πως οι παρατηρήσεις μας έχουν ληφθεί υπόψη και από, την άποψη, από τη δική μας άποψη μπορούμε να υποστηρίξουμε την προσέγγιση της Κομισιόν στο θέμα αυτό. Ποιος θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση και καταστροφή αγαθών που, παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα οι μεταφορείς έχουν τις πληροφορίες για τα, τα αγαθά που θα μεταφερθούν. Συχνά οι μεταφορείς ποτέ δεν βλέπουν ακριβώς τα ίδια τα αγαθά, αλλά βασίζονται στις πληροφορίες που τους δίνονται από τον ε, εξαγωγέ ή τον εισαγωγέα. Τώρα, η τον εισαγωγε τωρα η νομιμοτητα της εν λόγω πώλησης είναι θέμα, είναι αρμοδιότητα των τελωνιακών αρχών που εργάζονται με βάση τις αρχές που ισχύουν ή από τον ίδιο τον δικαιούχο του δικαιώματος αυτού πνευματικής ιδιοκτησίας, ο οποίος συχνά είναι ο μόνος που μπορεί να επιβεβαιώσει την ομιμότητα της συναλλαγής. Συχνά οι μεταφορείς ή άλλοι προμηθευτές υπηρεσιών πρέπει να ενημερωθούν από τον πελάτη για να μπορέσουν να αξιολογήσουν τον κίνδυνο και θεωρούμε πως αυτό είναι πολύ σημαντικό έργο και πολύ σημαντική συμβολή. Αξιολόγηση κινδύνου γίνεται από την, το ίδιο το τελωνίο και μπορεί να ε, σημαίνει κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες που απορρέουν και τις οποίες ορίζει το τελωνίο. Ο μεταφορέας εκτελεί αυτές τις αποφάσεις του τελωνίου, αλλά δεν μπορεί να τις λάβει τις αποφάσεις αυτές στη θέση του τελωνίου, των τελωνιακών αρχών. Ακόμα και αν ελέγξει τις, ε, τα αγαθά, θα, δεν μπορεί να γνωρίζει, ούτε μπορεί να, να ε, κατηγορηθεί ότι γνώριζε ή όχι την αυθεντικότητα αυτών των αγαθών. Επίσης, δεν θα πρέπει να κατηγορηθούν για την ρήξη μιας σύμβασης για την οποία δεν είναι υπεύθυνη για την ε, παραβίαση ή τη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας εφόσον αυτό δεν εμπίπτει μέσα στις δικές τους αρμοδιότητες. Ποιος ωφελείται τώρα από την παρακράτηση ή καταστροφή των ε, κατασκευθέντων προϊόντων. Αν τα αγαθά αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή απειλούν να υποβαθμίσουν τη συλλογή ε, φόρων και δασμών, είναι προς το δημόσιο συμφέρον να κατάσχονται ή να καταστρέφονται τα δημόσια αυτά αγαθά. Αν η κατάσχεση και η καταστροφή αυτών αγαθών εμπίπτει περισσότερο, στο, μάλλον βαραίνει τον ίδιο τον δικαιούχο, τότε είναι προς το συμφέρον του ίδιου του δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων να καταστραφούν αυτά τα αγαθά. Τα κόστη ε, τα φέρει ο δημόσιος τομέας είτε ο δικαιούχος ο οποίος θα πρέπει φυσικά όπου δει να ζητήσει αποζημίωση από τους ε, δράστες της παράνομης αυτής συναλλαγής. Συμπέρασμα. Οι μεταφορείς ή οι άλλοι προμηθευτές ε, τέτοιου είδους υπηρεσιών δυστυχώς δεν είναι σε θέση να ελέγξουν την αυθεντικότητα των προϊόντων που μεταφέρουν δεν έχουν περιθώρια λιγμού όταν ε, προκύπτει νέος, νέο κόστος υπό τη μορφή αποθήκευσης ή καταστροφής των αγαθών. Εν γέννη δεν μπορούν να ελέγξουν τα αγαθά τα ίδια καθώς οι συμβάσεις δεν επιτρέπουν το άνοιγμα πακέτων. Λαμβάνουν πληροφορίες που είναι πολύ σημαντικές για την ανάλυση κινδύνου και για τη διαχείριση του κινδύνου, αλλά οι πληροφορίες αυτές δεν επιτρέπουν καμία ε, ε, επιλογή ή άποψη να προκύψει για όσον αφορά τα αγαθά και την πιθανότητα αυτών να παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα. Επίσης δεν μπορούν, δεν είναι νομικά εξουδοτημένοι να αναγνωρίζουν την αυθεντικότητα των αγαθών και ούτε μπορούν να προβούν σε ανάλυση κινδύνου οι προμηθευτές υπηρεσιών. Δεν λαμβάνουν ωφέλη για την κατάσχεση, αποθήκευση ή καταστροφή παραποιημένων ή πλαστών ε, αγαθών οι μεταφορείς καθώς και οι προμηθευτές υπηρεσιών υλικοτεχνικών παρέχουν όσα στοιχεία τους ζητούνται. Και αυτό το κάνουν γνωρίζοντας ότι αυτή, αυτά τα στοιχεία είναι πολύ σημαντικά για τις σωστές διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου. Επίσης προσπαθούν να συνεργαστούν με τα ιστελωνιακές αρχές και άλλες αρχές στον μέγιστο δυνατό βαθμό προς όφελος ε, όλων. Ο κύριος Νιούμαν αναφέρθηκε στην σημασία της συνεργασίας με τα τελωνία που βασίζεται στην εμπιστοσύνη εκεί όπου μοιραζόμαστε πολύτιμες πληροφορίες και συμφωνώ απόλυτα με αυτήν την άποψη. Ωστόσο, η παροχή στοιχείων και η συνεργασία σε κάποια δομή με τα ιστελονικές αρχές και άλλες αρχές όσον αφορά τους ίδιους τους, φορεί, τους μεταφορείς ε, είναι σωστή, αλλά το να συμμετέχουν, να εμπλακούν περισσότερο πέρα δηλαδή από την ε, κανονική ε, ενημέρωση για την προστασία του δημοσίου ή να αναλάβουν την ευθύνη για μια ιδιωτική σύμβαση της οποίας δεν είναι συμβαλόμενα μέρη δεν είναι λογικό ούτε νομικά βάσιμο. Ε, δεν είμαστε λοιπόν μέρος ε, εμείς αυτής της διαδικασίας, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι η ευθύνη για το κόστος που σχετίζεται με την ε, αξιολόγηση και την επαλήθευση των παραβίασης ή μη των πνευματικών δικαιωμάτων. Και ως προς αυτή την πτυχή μπορούμε να υποστηρίξουμε και πάλι την πρόταση της Κομισιόν. Αυτά και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ και εγώ. Τελείωσε. Τελειώνει μάλλον ο πρώτος γύρος. Τελευταίος ομιλητής ο κύριος Στάλα από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών. Είναι το ανώτατο στέλεχος υπεύθυνο για την ανάλυση κινδύνου. Πραγματικός πρακτικός. Και θα μας μιλήσετε για την εφαρμογή, την προστασία μάλλον των πνευματικών δικαιωμάτων από τα γερμανικά τελωνία. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω εδώ σήμερα. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, όπως είπε ο κ. Κρόιτσμαν εισαγωγικά, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ είναι ότι είναι τεχνικός πολύ ο κανονισμός. Γι' αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στο ρόλο της δίκησης σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση των, ε, της παραποίησης. Θα ήθελα να κοιτάξουμε το τι κάνουμε σήμερα και μετά να αναφερθώ στη νέο κανονισμό που μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που είναι τα δυνατά και τα δύναμα σημεία. Θεωρώ ότι σημαντικό είναι ότι θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι συζητάμε ένα κανονισμό ο οποίος ε, αφορά ε, τα παραποιημένα προϊόντα. Δεν μιλάμε για μια νομοθεσία που αφορά προϊόντα που δεν πληρούν τις ε, προδιαγραφές ασφαλείας και το καθεξής. Υπάρχουν πολλές παραποίησεις που έχουν να κάνουν με παραποίηση δικαιωμάτων, οι οποίες κατεπιστάνονται με βάση τις εθνικές και κοινωτικές ε, αρχές. Η νομοθεσία μιλάει μόνο για τα πνευματικά δικαιώματα. Άρα, εδώ ο δικαιούχος αναφέρεται στις τελωνιακές αρχές όταν ανακαλύπτονται προϊόντα τα οποία ενδεχομένως να παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τότε θα προβούμε σε κατάσχεση των προϊόντων αυτών και μετά μέσω αστικής ευθύνης θα διευκρινιστούν κατά πόσον αποτελούν τα προϊόντα αυτά παραβίαση της νομοθεσίας και στην περίπτωση αυτή θα προβούμε σε καταστροφή των προϊόντων αυτών ή θα εκδικαστεί η περαιτέρω μεταχείριση των προϊόντων. Η τελωνιακή αρχή είναι τρίτο μέρος και μόνο σε αυτή τη διαδικασία. Όταν ο δικαιούχο και ο ιδιοκτήτης δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία, η τελωνιακή υπηρεσία απελευθερώνει τα προϊόντα αυτά. Και εδώ είναι η μεγάλη διαφορά με τις άλλες περιπτώσεις. Εδώ λοιπόν υπάρχει νομική σχέση μεταξύ, κατά την οποία μάλλον παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η τελωνιακή αρχή, η οποία όμως δεν θα πρέπει να μπερδευτεί με τα εθνικά μέτρα. Θα πρέπει να κοιτάξουμε το χρονοδιάγραμμα στα 15 χρόνια με τα οποία, στα οποία ασχολούμαστε με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδιαίτερα πέρσι, ήταν τεράστια η αύξηση των περιπτώσεων παραβιάσεων των πνευματικών δικαιωμάτων. Είναι σημαντικό όμω να διευκρινίσουμε τι κρύβεται πίσω από τι υποθέσει αυτέ. Κοιτώντα τα στατιστικά στοιχεία, διαπιστώνουμε ότι τα δέματα τα οποία περιλαμβάνουν πάνω από τρία προϊόντα αποτελούν 17% των ε, παραβιώσεων και 19% των ε, προϊόντων που κατασχέσαμε, δηλαδή μεγάλο ποσοστό των ε, δεμάτων, δεν περιλαμβάνει σχεδόν κανένα εμπόρευμα ή πολύ λίγα εμπορεύματα. Παρ' όλα αυτά, σημαντικό μέρος της εργασίας των τελωνίων ε, συνεπάγονται αυτά τα δέματα και για προσωπικό και για άλλα ζητήματα. Και τι κρύβεται πίσω από αυτά, το είπε ο κύριος Τσίμερμαν στην αρχή, ο 23% όλων των κατασχέσεων το 2010 ε, έγιναν στον ταχυδρομικό τομέα. Θα ήθελα ωστόσο να επιστήσω την προσοχή σας στις ποσοστώσεις σε ό,τι αφορά και τις οδικές μεταφορές και τις μεταφορές μέσω της θάλασσας. Ενώ ε, ο ταχυδρομικός κλάδος ε, ευθύνεται για το 23% αναφέρεται σε 5% των περιπτώσεων, ενώ 33% μεταφέρονται για θάλασσα και 51% μέσω οδικών οδών. 5% λοιπόν ταχυδρομικό κλάδο, περιφερειακό ποσοστό. Τα βασικά προβλήματα είναι στις μεταφορές ε, τις και τις θαλάσσιες. Αυτό τι σημαίνει ότι ταχυδρομικός κλάδος ε, ε, αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο ποσοστό του άχθους, αλλά δεν αποτελεί το σημείο εστίασής μας σε ό,τι αφορά ε, το, την αξία που εκπροσωπεί. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα προϊόντα εκείνα, τα οποία είναι τα πιο σημαντικά για την προστασία της ευρωπαϊκής έδρας. Και αυτό δεν είναι ο τομέας των ταχυδρομικών μεταφορών. Θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό. Και αυτά είναι τα βασικά σημεία στα οποία δραστηριοποιούμαστε. Χρησιμοποιούμε απλές διαδικασίες καταστροφής. Ε, πάνω από 21.307 περιπτώσεις είχαμε απλές καταστροφές και έτσι ε, πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά ε, ικανοποιήσαμε τα δικαιώματα των δικαιούχων σε ό,τι αφορά τις αστικές υποθέσεις παρουσιάστηκαν 70 72 εξ αυτών στη Γερμανία. Πολύ λίγες. Και αυτό μας οδηγεί στο επόμενο πρόβλημα, ότι δηλαδή έχουμε περίπου 1170 περιπτώσεις όπου ως τελωνίο θεωρήσαμε ότι είχαμε παραποιημένα προϊόντα και τελικά μετά από έλεγχος προέκυψε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν ε, ε, αυθεντικά τα προϊόντα, μη παραποιημένα. Και αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα μικρά πακέτα. Αν η ευθύνη για την απόφαση κατά πόσον πρόκειται για παραποιημένο ή μη προϊόν ε, ε, εμπίπτει και θα πρέπει να εμπίπτει στα τελωνία. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη, γιατί δεν έχουμε τι πληροφορίε για να αποφασίσουμε κατά πόσο πρόκειται για πραγματικό ή μη πραγματικό προϊόν. Ο μοναδικό που μπορεί να το κάνει αυτό είναι ο δικαιούχο, ο οποίο ωστόσο χρειάζεται να διαθέτει πολύ πιο εκτενείς πληροφορίες. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, και το είπα και εισαγωγικά, είναι ότι είμαστε ουσιαστικά τρίτο μέρος στην διαδικασία αυτή. Έχουμε στη Γερμανία 21.307 ε, περιπτώσεις το 50% των δικαιούχων δεν απάντησαν στις εκκλήσεις μας. Γιατί και έτσι, παρά τις προσπάθειες των τελωνίων, αναγκαστήκαμε να αφήσουμε ελεύθερα στην αγορά 1160 προϊόντα, παρόλο που είχε γίνει σχετική έρευνα, επειδή ο δικαιούχος δεν θέλει να αναλάβει το κόστος μιας ε, αστικής διοικής. Όσο υπάρχει λοιπόν σε πολλές περιπτώσεις που μπορεί ο δικαιούχος να λάβει ο ίδιος την προστασία του, δεν βλέπουμε την προστατιαξία αξία των τελωνίων. Θα θέλαμε να ε, δημιουργηθούν στενές σχέσεις συνεργασίας. Αυτό είναι πιο σημαντικό από κάθε νέα νομοθεσία για την καταπολέμηση παραβιάσεων των πνευματικών δικαιωμάτων για να εξαγάγουμε ένα συμπέρασμα. Τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε λύσεις αποτελεσματικές, όχι μόνο για τους δικαιούχους, αλλά δεδομένων των περιορισμένων πόρων και για την τελωνιακή αρχή. Τι σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μια τυποποιημένη προσέγγιση για όλα τα είδη των παραβιάσεων πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν υποστηρίζουμε την πρόταση να γίνει διάκριση μεταξύ ε, ευρεσιτεχνιών και λοιπόν δικαιωμάτων πνευματικής συντεκτησίας, γιατί σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποφασίσει το τέλειο τελικά αν ε, ε, ένα προϊόν αποτελεί ή μη παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Θέλουμε μία λύση η οποία θα δίνει μία σαφή λύση και μία σαφή διαπαφή στο τελωνία για να λάβει την απόφαση που πρέπει να προβεί η μη σε καταστροφή, γιατί μία διάκριση θα σήμαινε σημαντικές δυσκολίες για μας και θα μας οδηγούσε σαφώς σε ε, ζημία. Θα πρέπει επίσης να μην... θα έπρεπε να αποφύγουμε όλα τα βήματα τα οποία δεν είναι απολύτως απαραίτητα και σε αυτά συγκαταλέγεται και μία ενδιάμεση διαδικασία. τα οποία θα συνεπάγονταν και υπερβολικό άχθος. Επίσης, η γενικότερη προσέγγιση σε άλλους ε, τομείς ε, θέλουμε τήρηση των ε, διατάξεων ασφαλείας και θα πρέπει να διευκρινίζεται κατά πόσο τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν ήταν ημίδικε δικαιολογημένα. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε σαφή κατανομή των ε, ευθυνών, γιατί τα τελωνία είναι ε, ουδέτερο μέρο στη διαδικασία. Σε καμία φάση δεν θα μπορέσουμε να αποφασίσουμε αν πρόκειται για παραβίαση ή μη και κατά πόσον θα πρέπει να προβούμε ή όχι σε καταστροφή. Αυτά που προκύπτουν από το άρθρο 24 σε ό,τι αφορά τα μικρά δέματα, παρά το γεγονός ότι προκαλούνται μικρά προβλήματα, ε, ευθύνη θα πρέπει να παραμείνει στον δικαιούχο και αυτός είναι υπεύθυνο για την ανάληψη του κόστους. Και στη συνέχεια μπορεί μέσω δικαστικών αγωγών να ζητήσει αποζημίωση για τα έξοδα αυτά. Δύο σημεία ακόμα θα πρέπει να περιοριστούμε στις σημαντικές περιπτώσεις, στις οδικές μεταφορές, τις ε, θαλάσσιες μεταφορές και θα πρέπει να κοιτάξουμε και να λύσουμε το ζήτημα των ταχυδρομικών δεμάτων στην πηγή τους τα καταστήματα μέσω διαδικτύου, τα οποία θα πρέπει να φροντίσουμε να παρελιστούν, γιατί δεν μπορούμε να ελέγχουμε τόσο μεγάλο όγκο αποστολών κάθε χρόνο. Σας ευχαριστώ. Well, thank you very much for... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ πρακτική περιγραφή δεδομένων. Νομίζω ότι Όλες οι μαρτυρίες ήταν πάρα πολύ χρήσιμες και επέσυραν την προσοχή μας στα μικρά δέματα και τις επιχειρήσεις γύρω από αυτά. Και βεβαίως πολύ σωστά είπατε ότι δεν μπορείτε να διαμασολαβήσετε μεταξύ δέσμευσης κατάσχεσης και τα λοιπά. Είναι θέμα νομοθετικό. Συνάδελφοι, μπορείτε να πάρετε το λόγο για ερωτήσεις ή σχόλια. Ποιοι θα θέλουν να πάρουν το λόγο. Ο κύριος Κρόιτσμαν ξεκινάει και θα δούμε αν υπάρχουν άλλες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Τιμπέρ μας ανέφερε ότι μεταφορείς οι οποίοι κάνουν μια παράδοση δεν ε, αισθάνονται υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των ε, ε, πορευμάτων. Συναντήθηκα πρόσφατα με έναν δικαιούχο, ο οποίος μας ανέφερε ότι παραποιημένα προϊόντα παραδόθηκαν από την Κίνα και υπήρχε ευκαιρία να καταστραφούν τα εμπορεύματα αυτά. Καταστράφηκαν λοιπόν και στη συνέχεια προσπάθησαν να αποζημιωθούν για το κόστος αυτό, αλλά δεν υπήρχε καν ο δηλωμένος αποστολέας. Και τώρα ερχόμαστε κύριε Στόλεφ, στην ερώτηση την οποία αναφέρεται στο θέμα που αναφέρατε για τις θαλάσσιες μεταφορές. Στις ταχυδρομικές ε, αποστολές καταλαβαίνουμε τι λέτε. Αλλά αν ένας πλειοκτήτης ε, μεταφέρει από μία χώρα σε μία άλλη χώρα μεγάλα κοντέινερ και στη συνέχεια αποδεχτεί ότι δεν υπάρχει ο αποστολέας και ο πληκτήτης ε, δηλώσει ότι α, λυπάμαι, τι να κάνουμε. Εσείς ε, το ελέγχετε αυτό. Εγώ προσωπικά λοιπόν έχω πρόβλημα γιατί δεν μιλάμε για μικροποσότητες, μιλάμε για ολόκληρα κοντέινερ, ολόκληρα βότια. Πώς μπορούμε λοιπόν να καταστήσουμε υπεύθυνους και τους πλειοκτήτες Θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη. Να μου πείτε επίσης ο κύριος Στόλε, αν σωστά κατάλαβα, θεωρείτε ότι δεν είναι σκόπιμη μία ακρόαση. Τι θα γίνει, ο δικαιούχος λέει προφανώς ότι θα πρέπει να καταστραφεί το προϊόν και λέτε εσείς ότι δεν υπάρχει νόημα. Πώς θα ε, λυθεί το πρόβλημα αυτό όμως. Thank you. I think Ευχαριστώ. Πολύ σημαντικά ζήτηματα. Μου έχει εντυπωσιάσει το σχόλιο του κυρίου Στόλερ, το οποίο σχετίζεται με αυτό που είπε ο εισηγητής, την αδράνεια δηλαδή των δικαιούχων. Ε, έχω εργαστεί και εγώ σε αυτόν τον τομέα με την Γενική Διεύθυνση Ταξούτ και πράγματι φαίνεται να υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου δικαιούχοι αυτοί ε, δεν είναι καθόλου πρόθυμοι να εμπλακούν στην διαδικασία να προασπίσουν τα σήματά τους. Και ο κύριος Μιούλερ είναι ο βασικός εκπρόσωπος αυτού του χώρου. Θα ήταν ενδιαφέρον να μας πείτε αν δεν εμπλέκονται διότι οι διαδικασίες είναι πολύ περίπλοκες και η πρόταση κάπως διευκολύνει τις διαδικασίες για να υποστηρίξουν τα δικαιώματά τους, αλλά είναι διατεθειμένοι να εμπλακούν και να φέρουν και το κόστος της καταστροφής των προϊόντων, των παραποιημένων βεβαίω. Να ρωτιέμαι. Άλλος συνάδελφος, ο κύριος Καρίδα. Κύριο κύριος μάλλον. Έχω ένα ε, ερώτημα για το άρθρο 4. Δεν ξέρω αν είναι ο κατάλληλη στιγμή να το θέσω ή στην επόμενη σύνοδο. Θα σας δώσω το λόγο στον επόμενο γύρο. Ναι, νομίζω ότι είναι καλύτερα για το άρθρο 4. Ο επόμενος γύρος. Κυρία Γκάλο τώρα. Κύριε Πρόεδρε, Άκουσα και τους τέσσερις παρεμβαίνοντες. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν ουσιαστικά προβλήματα ενημέρωσης για τις τελωνιακές υπηρεσίες. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η στιγμή, αλλά έχω μία ερώτηση για το τελευταίο άρθρο της πρότασης. Ανταλλαγή στοιχείων, δεδομένων μάλλον, γιατί μου φαίνεται ότι η πρόταση της Κομισιόν δεν είναι επαρκής θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε την άποψη των εμπειρογνωμόνων μας σχετικά με το πώς θα μπορούσε να συσταθεί μια βάση δεδομένων που είναι το και το κλειδί μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον που ζούμε. Είναι εργαλείο, εργαλείο αποτελεσματικότητας για την νομοθεσία μας στην εκεί. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ποιος θα ήθελε από τους εμπειρογνώμονές μας να, μας, να σχολιάσει. κύριος Ζήμερμαν. Μετά ο κύριος Νιούμαν. Νομίζω ότι και ε, το έχετε καλύψει και οι τέσσερις. Απλώς κάντε μας ένα σύντομο σχόλιο στο ζήτημα που τίθηκε. Κύριε Ζήμερμαν, έχετε κάποιο σχόλιο σε σχέση με τα σχόλια που γίνανε. Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε. μία δράνεια των δικαιούχων. Πάρτε τον αριθμό των αιτήσεων παρέμβασης που έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει κινητοποίηση των δικαιούχων. Από μερικές χιλιάδες, τώρα έχουμε περάσει στις 16.000 νομίζω. Λοιπόν, υπάρχει κινητοποίηση των δικαιούχων του Το θέμα, το πρόβλημα είναι το, τα τα ταχυδρομικά δέματα, διότι αν ε, επιδιώξουν μια προσφυγή για τα 3, 5, 6 προϊόντα, ε, προσλάβουν δικηγόρο κτλ. Αυτό θα τους στοιχήσει πολλαπλάσια από τα παραποιημένα. Αυτό είναι δεδομένο. Στο παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει κινητοποίηση των δικαιούχων σημάτων, ακόμη και αν καμιά φορά Υπάρχουν ορισμένες αντιπαθητικές ε, τακτικές που τα βρίσκει ο Αποστολέας με ε, και ρυθμίζονται τα ζητήματα. Στο περιθώριο βέβαια. τώρα, όσον αφορά τη βάση των δεδομένων. Πολύ σημαντικό θέμα. Δεν είμαστε ειδικοί για να κρίνουμε αυτό το άρθρο. Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι στο επίπεδο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Τελωνίων. Έχουμε μία βάση δεδομένων, την EPM, που δεν ποσοτοποιεί, ποσοτικοποιεί ε, τα δεδομένα αν θέλετε, αλλά δίνει τη δυνατότητα στον τελωνιακό να ανοιχνεύσει το πλαστό από το αληθινό. Γιατί ότι έχουμε ψευδοποιότητα, αν θέλετε. Είναι, υπάρχει δυσκολία για το τελωνιακό να διαπιστώσει αν είναι πλαστό ή γνήσιο. Ε, οι περισσότεροι δεν μπορούν να διαχωρίσουν. Καμιά φορά χρειάζομαστε χημικές αναλύσεις για τα προϊόντα για να διαπιστώσουμε αν είναι πλαστό απομίμηση δηλαδή γνήσιο. Και είναι δύσκολο ο τελωνιακός να αποφασίσει. Οπότε η Παγκόσμια Οργάνωση Τελωνίου ξεκίνησε μία βάση δεδομένων που θα επιτρέψει σε αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη σειρά να έχουν πλήρη ενημέρωση για να ξεχωρίσουν το γνήσιο από, την απομίμηση. Ο κύριος Νιούμαν τώρα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα απαντήσω σε δύο από τα ερωτήματα αδράνεια των δικαιούχων. Σε συνέχεια, από όσα είπε ο κύριος Ζήμερμαν, και εγώ επιβεβαιώνω ότι έχει υπάρξει μεγάλη ε, ενεργοποίηση της βιομηχανίας των τελευταία 5 με 10 χρόνια. Βεβαίω δεν μπορώ να ε, δικαιολογήσω την αδράνεια σε εξατομικευμένες περιπτώσεις. Χρειάζεται κανείς να ξέρει και τις λεπτομέρειες βεβαίως για να καταλάβει καλύτερα την αδράνεια μπορώ να πω ότι τα μέλη της ITA πραγματικά έχουν ε, συνέστηση αυτού του θέματος και είναι υπεύθυνοι πολιτές. Τώρα, όσον αφορά τα, την πληροφόρηση που είναι θέμα κλειδί, οπωσδήποτε ε, δεχόμαστε να είμαστε υπεύθυνοι κάτω από ορισμένε συνθήκες, αλλά όταν είμαστε, έχουμε τα χέρια δεμένοι δεμένα και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που λάβαμε για να πάμε στην πηγή, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ ε, εκνευριστικό να εμπλακεί κανείς στη διαδικασία η οποία μόνο καταστρέφει τα προϊόντα. Ενδιάμεση τώρα. Πιστεύω ότι εδώ η μεγαλύτερη ανησυχία μας είναι να μην μεταφέρουμε το κόστος σε οποιονδήποτε ενδιάμεσο είναι διαθέσιμος. Θέλουμε να αναζητηθεί η ευθύνη, η πραγματική για την υπόθεση και αυτή η ευθύνη ε, σημαίνει ότι πρέπει να ξέρουμε καλύτερα τον πελάτη. Ε, χρειαζόμαστε τη δέουσα επιμέλεια, ώστε όταν ο δικαιούχος να μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για να επιτύχει και αποζημίωση. Να υπάρχει τουλάχιστον η, ε, η πιθανότητα να έχουν συλλεγεί πληροφορίες κάπου, ξεκινώντας. Ο κύριος Βαντεμπέρ τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Κρόιτσμαν για την ερώτησή σας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και επίκαιρη. Συνήθως οι μεταφορείς πάντα τα γνωρίζουν αυτούς με τους οποίους έχουν ένα συμβόλαιο. Λοιπόν, αν έχουν ένα συμβόλαιο με τον φορτωτή, με τον αποστολέα, θα τον γνωρίζουν. Και αυτός και θα τους πληρώσει. Συνεπώς είναι γνωστός. Στις εμπορικές συναλλαγές βεβαίως εμπλεκόνται πολλά μέρη. Και αν το μέρος που διατάσσει τη μεταφορά, την παροχή δηλαδή υπηρεσιών από τον μεταφορέα. Δεν είναι αυτός αλλά ο αποστολέας, αλλά ο παραλήπτης, τότε μπορεί αυτός να μην είναι γνωστός από τον μεταφορέα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ήταν καλή πρακτική ε, να ήταν γνωστός και αυτός. Ένας προθητής μεταφορών πρέπει να γνωρίζει βεβαίως το, στον εφικτό βαθμό του συναλλασσόμενους μαζί του. Υπάρχει και ένα πρόγραμμα AO στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ένας από τους όρους για να επιτύχει κανείς αυτό το... την πιστοποίηση αν θέλετε. Ακριβώς εξασφαλίζει ότι γνωρίζει τους εμπορικά συναλλασσόμενους μαζί του. Είναι θέμα ποιότητας της υπηρεσίας, συμφωνώ. Αλλά δεν μπορεί να αποτελεί γενική προδιαγραφή και να συνεπάγεται γενικό επιμερισμό του κόστους δέσμευσης, αποθήκευσης ή καταστροφής. Είναι διαφορετικό το ζήτημα εδώ. Η πιστοποίηση αυτή εννοώ. Ποιος είναι τώρα αυτός ο οποίος υποφελείται από αυτή την ενέργεια την τελωνιακή. Βεβαίως το κοινό πρώτα απ' όλα ε, όσον αφορά την ασφάλεια και βεβαίως και ο δικαιούχος του σήματος. Ο μεταφορέας δεν έχει κανένα όφελος και ουσιαστικά δεν έχει και τη δυνατότητα να παρέμβει στις περισσότερες περιπτώσεις. Όταν πρόκειται για δέουσα επιμέλεια ή ποιότητα υπηρεσιών, ε, συμφωνώ ότι προσπιζόμαστε την προώθηση αυτών των αξιών. Ακριβώς για να υπάρχει αυτή η πιστοποίηση. Ο κύριος Τάλε. Σας ευχαριστώ για να συμφωνήσω ότι και η ποιότητα των δεδομένων είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για τις τελωνιακές αρχές, γιατί όπως αναφέρθηκε προηγουμένως ε, βασιζόμαστε σε μια προσέγγιση βάσει αξιολόγησης κινδύνου. Άρα είναι σημαντικό να ξέρουμε ποιο στέλνει και ποιο παραλαμβάνει ένα δέμα, προκειμένου να ε, εντοπίζουμε τα παραπημένα προϊόντα στο βαθμό του δυνατού. Άρα υποστηρίζουμε σαφώς την προσέγγιση για την βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων. Για να απαντήσω στην ερώτησή σας κύριε Κρόιτσμαν για το ποια διαδικασία θα θέλαμε να προτείνουμε και ποια διαδικασία εφαρμόζουμε χωρίς μεγάλα προβλήματα, χωρίς ε, ουσιαστικά προβλήματα στην πράξη, επικοινωνούμε με τους δικαιούχους, τους ενημερώνουμε για μια ενδεχόμενη ε, αποστολή που έχει παραβιάσει τα πνευματικά της δικαιώματα και στη συνέχεια ο δικαιούχος ε, μας αποστέλνει μία γραπτή δήλωση για την απλοποιημένη καταστροφή των προϊόντων. Αυτό στην πράξη δεν παρουσιάζει προβλήματα. Στην αρχή ίσως είχε παρουσιάσει κάποια προβλήματα γιατί δεν λαμβάναμε γραπτή δήλωση, αλλά με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε ότι λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα ε, του καθενός γιατί τηρούνται οι προθεσμίες και επίσης σε περίπτωση δικαιούχων όπου υπάρχει κίνδυνος να γίνει κατάχρηση της διαδικασίας, ε, ασφαλώς ε, ζητούμε σχετική συνεργασία. Είναι αποτελεσματική λοιπόν και γρήγορη αυτή η διαδικασία και έτσι αποφεύγεται ε, η επιβάρυνση του δικαιούχου αλλά αυτό που παραμένει είναι ότι το άτομο στο οποίο, με το οποίο η επικοινωνεί η τελωνιακή αρχή θα πρέπει να επικοινωνεί με τις τελωνιακέ αρχές για ενδεχόμενο ε, δικαστική αγωγή. Το θέμα για την κυρία Γκάλα, το θέμα είναι πώς μπορούμε τις διάφορες ε, βάσεις δεδομένων που υφίστανται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, να τις συμπληρώσουμε τη μία με την άλλη. Έχουμε μία βάση δεδομένων στη Γερμανία που συμπεριλαμβάνει ε, δεδομένα από όλη την Ευρώπη και χρησιμοποιούμε ε, διάφορα δεδομένα από διάφορες ενώσεις και θέλουμε στο μέλλον να συνεργαζόμαστε και με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο κατά της πειρατείας εμπορευμάτων, με το οποίο συνεργαζόμαστε στενά. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες ε, ε, συνδέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πρόβλημα είναι να εφαρμοστούν αυτά τα στοιχεία τα οποία μας μεταβιβάζονται και βλέπουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι ελάχιστες οι πληροφορίες που μας χορηγούν οι δικαιούχοι για την προστασία των προϊόντων τους, γιατί πολύ απλά φοβούνται ότι θα δημοσιευτούν αυτά τα στοιχεία και θα είναι πολύ πιο εύκολο για τους ε, υπεύθυνου τη παραποίηση να κάνουν άλλη παραποίηση. Εμεί όμω δεν έχουμε δυνατότητα να διαπιστώσουμε κατά πίσω πρόκειται για παραποίηση ή όχι. Θα θέλαμε λοιπόν όχι απαραίτητα μία νέα βάση δεδομένου αλλά μία πιο στενή ανταλλαγή στοιχείων και ε, μία κάλυψη ως προς το απόρριτο. Μία έκκληση. Αν ένας δικαιούχος θεωρεί ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει μια δικαστική αγωγή για δύο-τρία προϊόντα, μπορεί να καταθέσει μια αίτηση. Το οποίο επιβαρύνει τον φορολογούμενο σε αντίθεση με τη μέθοδο αυτή, η οποία ουσιαστικά είναι πιο γρήγορη και οικονομική. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Ελπίζω να μπορέσετε να μείνετε μαζί μας για να έχουμε και ευκαιρία για περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων αργότερα. Θα περάσουμε τώρα στο δεύτερο γύρο που εξετάζει πιο συγκεκριμένα τον αντίκτυπο στους καταναλωτές ε, και βεβαίως θα καλυφθεί το θέμα των μικρών δεμάτων που αναφέρθηκε νωρίτερα ε, και καλωσορίζω την πρώτη μας ε, ομιλήτρια, την κυρία Κριστιαν Λάι ελπίζω να το προσφέρω σωστά, που είναι Γενικός Διευθυντής της Ένωσης ε, Κατασκευαστών. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, είναι τιμή μου που παίρνω το λόγο σήμερα εδώ και σας ευχαριστώ που καλέσατε την ε, ένωσή μας την UNIFAB. Η ένωση την οποία εγώ, της οποίας εγώ είμαι διευθύντρια έχει 200 μέλη που αντιπροσωπεύουν ε, τα πνευματικά δικαιώματα όλους τους βιομηχανικούς τομείς και που συνεργάζεται τακτικά με άλλες εθνικές ενώσεις για να προωθήσει την ανάπτυξη της ε, πνευματικής ιδιοκτησίας εξού και οι τακτικές εκστρατείες, η επικοινωνία ε, με το ευρύ κοινό και η εκστρατεία του 2010 επέτρεψε σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιήσουν το ίδιο σύνθημα ή σλόγγαν προς τον καταναλωτή τέλος στα παραποιημένα. Ε, είμαστε λοιπόν ε, θεωρούμε μάλλον ως μια ευκαιρία ε, τον ε, προτινόμενο κανονισμό για εξυγχρονισμένα ε, μέσα που θα δοθούν στον, τα, στα τελωνιακές αρχές έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί ένα φαινόμενο που δεν σταματά να αυξάνεται ώστε να μπορέσει να αναπτύσσεται για να μπει μέσα στο νόμιμο εμπόριο χρησιμοποιώντας όλα τα όρια των σημερινών ισχύουσεων διατάξεων και βεβαίως την μη προσαρμογή αυτών των διατάξεων στην κυβερνοπαραποίηση. Είναι έχουμε κάνει αυτή τη διαπίστωση και το διαπιστώνουν και καθημερινά οι επιχειρήσεις μας που ασχολούνται με την καταπολέμηση των παραπημένων προϊόντων. Είμαστε πεπισμένοι ότι, έχω, ότι αν δοθούν στα τελωνία καλύτερα εργαλεία θα αντιμετωπίσουμε καλύτερα αυτό, αυτήν την πληγή. Έχουμε ένα συγγραφέα που πήρε το βραβείο Κονκούρου πέρυσι που, ονομάζεται Μισελ Ουελμπέκ και είχε γράψει ένα βιβλίο που ονομάζεται «Οι δυνατότητες ενός νησιού». Αυτό που περιμένουμε εμείς είναι οι, δυνα... δυνατότητες να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα. Δύο ιδέες για να σας αναφέρω κάποιες πιο τεχνικές σκέψεις. Η Ευρώπη πρέπει ενωμένη να σταθεί αν... εναντί των πλαστών αγαθών, γιατί ε, ε, είναι το αδύναμο στοιχείο ο έλεγχος στην Ευρώπη. Αν η Ευρώπη δεν θέλει να, να αποτελέσει μόνο το πεδίο διέλευσης των παραπημένων προϊόντων, θα πρέπει ενωμένα και εναρμονισμένα να αντιμετωπίσει τα παραπημένα προϊόντα που έρχονται εκτός κοινότητας. Ε, και αυτές οι δυνατότητες ελέγχου θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες τόσο από το καθεστώς της ταξιδιού όσο και από το είδος του δικαιώματος που έχει κλαπεί. Και γι' αυτό και προβλέπει η Κομισιόν αυτή τη δυνατότητα παρέμβασης για κάθε είδος δικαιώματος και γι' αυτό και χαιρετίζουμε αυτή την πρόταση. Θεωρούμε πως το μήνυμα που στέλνεται στο οργανωμένο έγκλημα από την Ευρώπη είναι πολύ ε, ισχυρό. Πιστεύουμε πως είναι σημαντικό να ελέγχεται αυτό που εμείς αποκαλούμε την ε, ε, τον εκφυλισμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όπως αυτά που ονομάζονται look-alike. Είναι δηλαδή αθέμητος ανταγωνισμός, άλλοι δεν το θεωρούν αυτό ε, πάντως πρόκειται για ένα είδος ε, που θέτει σε απόλυτη ανεξιοπιστία την εργασία των ευρεσιτεχνιών γιατί αυτά τα προϊόντα εκφυλίζουν τη φύση των πνευματικών δικαιωμάτων. Έπειτα, τμηματικές αποστολές. Ε, εδώ έχουμε απλά αποστολές που είναι κομμάτια προϊόντων παραποιημένων. Ορίστε. Κοιτάξτε. Φρίκι. Φρύ και για έναν δικαιούχο πνευματική ιδιοκτησία και για ένα τελωνιακό. Μπορεί να είναι ένα περαστικό, διέλευση. Δηλαδή, και αυτό βρέθηκε σε έναν επιβάτη μάλιστα, δεν έχει σχέση με έναν συμβατικό τουρίστα που επιστρέφει με τα σουβενίρ του. Εδώ είναι ένας επαγγελματία που είναι ένα από τα μυρμήγκια ενό μεγάλου δικτύου. Τι γίνεται λοιπόν μετά αρμολόγηση στην Ευρωπαϊκή Επικρότεια. Εδώ είναι ρολόγια αλλά και τα τηλέφωνα, τα φάρμακα, ε, τα ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς ε, και πιστεύουμε ακριβώς ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μορφή της παραποίησης, γιατί εν γέννη αυτά τα προϊόντα, αν τα δούμε μονομένα, είναι μικρής αξίας. Μάλιστα, χωρίς καμία εμπορική αξία μπορεί να θεωρήσει κανείς και πολύ συχνά αυτά τα προϊόντα ακριβώς ε, στέλνονται σε μικρά δέματα. Για τα παράλληλα δίκτυα τώρα να σας μιλήσω. Εδώ βρίσκουμε και πάλι η παραποίηση. Πιστεύουμε πως πρέπει να ελεγχθούν και επίσης η αρχή της περιφερειακής εξάντληση των πραγματικών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Αυτό ε, λειτουργήσε πάρα πολύ καλά όσον αφορά τον έλεγχο των ε, κρασιών και των αλκοολούχων ποτών και μάλιστα λειτουργήσε πάρα, καλά, πάρα πολύ καλά στα σύνορα με την ε, Ρωσία. Και μάλιστα η Ρωσία η ίδια έχει τώρα υιοθετήσει το ίδιο σύστημα ελέγχου. Α έρθουμε τώρα στα μικρά θέματα. Δεν θέλουμε εδώ να τιμωρήσουμε οποιοδήποτε προσωπικό μεμονωμένο μάλλον καταναλωτή. Αυτό το είδο αποστολής κρύβει ένα σωρό είδη που δεν έχουν καμία χρήση, καμία σχέση με, το, με, με, με την παραποίηση. Ο, ο έλεγχος προβλέπεται στο 24 της πρότασής σας και θεωρούμε πως είναι ιδιαίτερη η μεταχείριση που πρέπει να υπάρχει γιατί έχουμε 20% κατασχέσεις που αυτή τη στιγμή εντοπίζονται από, τις, από τα τελωνία και που είναι παραγγελίες μέσω ίντερνετ. Αυτή η παραποίηση επικίνδυνη πολύ συχνά στέλνεται με ένα απλό μια απλή επιστολή και είναι οι περίφημες πλακέτες φαρμάκων που παραγγέλνονται μέσω ίντερνετ. Και γνωρίζουμε πως τα μικρά δέματα είναι ένα μέτρο για τα δίκτυα να ελέγξουν την αντίδραση των τελωνιακών, να δουν αν γνωρίζουν αυτή τη νέα μορφή δηλαδή παραποίησης. Η ευκολία Αυτόν τον ελέγχουν ακριβώς γιατί ε, τα τελωνία είναι ένας πεπερασμένος αριθμός ε, υπαλλήλων και πρέπει να συνδέονται με, μια συγκεκριμένη απλοποιημένη διαδικασία με στόχο την απόσυρση του εμπορεύματος ώστε να μην μπει στα εμπορικά κυκλώματα και αυτό όσο γίνεται πιο σύντομα. Και αυτό το προβλέπει μάλιστα το άρθρο 24 και η πρόταση αυτή ε, κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να εγκριθεί γιατί είναι πολύ ρεαλιστική. Ε, αντίθετα θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε δύο θέματα. Τι σημαίνει μικρό ε, δέμα. Ο ίδιος ο τελωνιακός θα κρίνει αν το συγκεκριμένο δέμα είναι μικρό ή όχι. Αν πρόκειται για μια ε, παραγγελία μέσω ίντερνετ, πολλές φορές βλέπουμε ότι μπορεί να στείλουν παραποιημένες ε, τσάντες ε, Louis Vuitton ή Gucci ή ακόμα και απομιμήσεις παλτών Burberry και ούτω καθεξής. Είναι πολλές οι μάρκες, πολλά τα σήματα που κινδυνεύουν εδώ τι γίνεται αν τελικά αυτό το δεν θεωρηθεί μικρό δέμα. Και έπειτα αυτή η διαδικασία είναι τόσο απλοποιημένη που τελικά αφήνει απ' έξω τον δικαιούχο των πνευματικών δικαιωμάτων που δεν έχει λόγο, ούτε μπορεί να κάνει τίποτα, ούτε ενημερώνεται για τη διαδικασία. Και εδώ έχω την εντύπωση και συμφωνώ με τα όσα έλεγε ο εκπρόσωπο των Γερμανικών Τελωνίων, πω ε, πρόκειται λίγο να, ότι θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε και ότι όταν ε, ο δικαιούχο παρεμβαίνει, παρεμβαίνει μόνο για να κρίνει ως εμπειρογνώμονας του προϊόντος του ε, για να επιβεβαιώσει τις υποψίες των τελωνίων, των τελωνιακών αρχών. Αν κάνουμε κάτι τέτοιο θα έχουμε απλά τελωνιακούς που τι θα κάνουν, ήδη θα είναι μεγάλο πολύ, αλλά που εν πάση περιπτώσει θα πηγαίνουν προς τα παραπημένα προϊόντα που γνωρίζουν καλύτερα, αυτά που βρίσκονται στη βάση δεδομένων και εις βάρος μιας ενημέρωσης διαρκούς που αντίθετα τα δίκτυα των ε, παραχαρακτών δεν διστάζουν να κάνουν. Ο εντοπισμός λοιπόν θα πρέπει να γίνεται εγκαίρος. Δεύτερη ιδέα είναι ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να γίνει ένας χώρος διέλευσης των παραπημένων προϊόντων. Γιατί να ελέγξει κανείς τη διέλευση σημαίνει ότι τα παραποιημένα προϊόντα δεν φτάνουν στην Ευρώπη ακριβώς με μορφή μικρών δεμάτων και μέσω παραγγελιών στο ίντερνετ. Εάν αποφασίσουμε να ελέγξουμε το τράζιτ, τότε αναθέτουμε στους ε, τελωνιακούς να δείξουν από πριν ότι προβλέπεται επιστροφή στην Ευρώπη. Η διαφορετικά στόχευση με επιτόπου δεν θα είναι δυνατή και άρα άλλη μια φορά θα πρέπει να διακριθεί το, το καθεστώς του ταξιδιού του αγαθού από την ε, παραποίηση. Έχω την εντύπωση πως η Ευρώπη που ακόμα και σε οικονομική, περίοδο οικονομικής κρίσης και που είναι πιο τυχερή και πιο πλούσια από την Αφρική θα πρέπει να κάνει αυτό το έργο του φίλτρου από την Αφρική, την Ασία και στην Λατινική Αμερική επίσης, όπου δεν υπάρχει μόνο η Βραζιλία. Ε, πολύ συχνά να αναπαυόμαστε στις δάφνες μας, ενώ πολύ γρήγορα τα εμπορεύματα αυτά μπαίνουν στην αγορά. Έχουμε έλεγχο 50% του εξοκοινοτικού εμπορίου που έρχεται και μπαίνει στις αγορές και ίσως να μην πρέπει να αυξηθεί αυτό το ποσοστό. Η παραποίηση σημαίνει μεγάλη συνεργασία, στενή συνεργασία ανάμεσα στους δημόσιους, ε, στις δημόσια αρχές και τους εμπόρους. Η πρόταση του 19 ωστόσο δεν προβλέπει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί παρά μόνο για να ενεργήσουμε στην, ε, δικαστικά στη χώρα μας. Ο, η Ευρώπη μπορεί να στείλει ένα μήνυμα ισχυρό σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο λέγοντας ότι όταν βρίσκουμε κάτι το οποίο δεν είναι εξοκοινωτικό να επιτρέψουμε στο δικαιούχο να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να βρει την αλυσίδα του ε, εμπορίου και να μπορέσει έτσι να διαλύσει αυτή την αλυσίδα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συμβολή σας. Ήταν πραγματικά ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε όσον αφορά το θέμα των μικρών δωμάτων, δεμάτων με που χρησιμοποιούνται για παραβίαση του συστήματος και για την πρόθεση απομιμήσεων. Έχουμε τον Keith Warren τώρα. Είναι διαχειριστής τελωνιακός της UPS στην Ευρώπη. Είναι εμπειρογνώμονος σε αυτό το θέμα, πολύ δραστήριος. Keith, έχεις μόνο 10 λεπτά σε προειδοποιώ για να μας πεις λίγα πράγματα γύρω από τις εμπειρίες σου. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω λέγοντας ε, μάλλον θα σας δώσω ορισμένα στοιχεία για τη μεταφορά express. Πώς καταπολούμε τις απομιμήσεις και ε, πώς ανησυχούμε για την έλλειψη ορισμού των μικρών δεμάτων. Λυπάμαι για το μικρό μέγεθος των εικόνων στην οθόνη. Φαντάζομαι ότι αυτό οφείλεται στο μικρό, δεν οφείλεται στο μικρό αριθμό παραποιημένων που βρήκαμε. Εν πάση περιπτώσει, βασικά μεταφέρουμε από τη μία πόρτα στην άλλη ένα δέμα σε όλο τον πλανήτη. Αυτό που έχει συμβεί τα τελευταία 20-25 χρόνια είναι ότι οι επιχειρήσεις έχουν αλλάξει τον τρόπο που λειτουργούν και χρειάζονται ακριβίας υπηρεσίες. Είμαστε σημαντικοί λοιπόν και για την ε, εσωτερική αγορά και για το διεθνές εμπόριο. εμπόριο 30 εκατομμύρια φορτία έχουμε καθημερινά, 220 χώρες εξυπηρετούμε, 1.700 αεροπλάνα έχουμε, 200.000 οχήματα και βεβαίως κάνουμε πάρα πολλούς εκτελονισμούς. Ένα κομμάτι των εκτελονισμών συνεπάγεται ότι δίνουμε πληροφορίες εκ των προτέρων για όλα τα θέματα τα οποία διακινούμε. Από την άποψη των υπηρεσιών Express σημαίνει ότι μεταφέρουμε υψηλής εμπεστησίας φορτία μεγάλης αξίας και παρακολουθούμε το εμπόρευμα το οποίο μεταφέρουμε συνεχώς με υψηλή τεχνολογία. Έχουμε φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία μεταφέρουμε σημαντικά για κάθε τομέα. Υποστηρίζουμε έντονα την την προσέγγι... μια αποτελεσματική προσέγγιση καταπολέμησης με βάση την ανάλυση κινδύνου καταπολέμησης των απομιμήσεων. Με την ταχύτητα που μεταφέρονται σήμερα τα φορτία, μπορείτε να καταπολεμήσετε την απομίμηση μόνο με άριστη ανάλυση κινδύνου. Αν το εξασφαλίσουμε αυτό έτσι, θα μπορέσουμε να καλύψουμε το μεγαλύτερο όγκο των φορτίων, να κινούνται ελεύθερα αυτά και με ασφάλεια. Ιδιαίτερα την εποχή αυτή οι επιχειρήσεις μας στην Ευρώπη πρέπει να εισάγουν και να εξάγουν με ταχύτητα. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν σαν μεταφορείς. Και όταν λέω μεταφορείς μιλάω ακριβώς για υπηρεσίες express παρέχουμε πληροφορίες παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, σημάτων κτλ. Όταν μας το ζητούν οι διάφορες αρχές και σύμφωνα με το εφαρμόσιμο δίκαιο, εφαρμοστέο δίκαιο. Ε, ο έλεγχος διεύθυνσης παραλήπτη, η αποστολέα ή ο έλεγχος ε, χνηλάτιση του φορτίου. Αυτά πραγματοποιούνται όταν μας ζητούνται κατόπιν αίτησης δηλαδή, διότι δεν είμαστε εμείς ειδικοί επί των σημάτων ή των πνευματικών δικαιωμάτων. Η έλεγχη που κάνουμε είναι βασικά για την ασφάλεια των πτήσεων. Δηλαδή προστατεύουμε το αεροσκάφος το οποίο μεταφέρει και το πλήρωμα. Τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν είμαστε ειδικοί. 16 χρόνια υπηρέτησα στο τελωνίο, στα τελωνία. Έχω δει όλων των ειδών τα φορτία, αλλά η επιβεβαίωση και η συμμόρφωση με τα πνευματικά δικαιώματα δεν είναι δυνατόν να ε, πραγματοποιηθεί από τα τελωνία. Δεν, κανένας δεν είναι εξουσιοδοτημένος για να προσδιορίσει το φορτίο οι υπαλληλοί μας δεν πρέπει να προσδιορίζουν τις παραβιάσεις της νομοθεσίας. Είναι περίπλοκη αυτή η διαργασία. Τώρα, η πρόταση της Κομισιόν όσον αφορά τα μικρά δέματα δεν τα προσδιορίζει. Και από την άποψή μας αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο, διότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές παραπομπές στο δίκαιο, στα μικρά δέματα. Αλλά δεν υπάρχει ένας γενικός ορισμός αυτών των μικρών φορτίων ή δεμάτων. Οπωσδήποτε δεν υπάρχει στον εξυγχρονισμένο τελωνιακό κώδικα τέτοια, τέτοιος ορισμός και ξέρουμε πόσος χρόνος απαιτείται για την εφαρμογή του επικαιροποιημένου κώδικα. Ο τελωνιακός κώδικας σήμερα λέει προϊόντα και μικρά δέματα τα οποία πηγαίνουν από ιδιώτες σε ο ιδιώτη. Μικρό δέμα λοιπόν. Τώρα, η νομοθεσία η φορολογική αναφέρεται στα μικρά φορτία με τον ίδιο τρόπο Πάλι αναφέρεται δηλαδή σε ιδιώτη που αποστέλνει σε ιδιώτη σε άλλο κράτος μέλος. Δηλαδή η υφιστάμενη νομοθεσία δεν μας βοηθάει καθόλου σχετικά με τον ορισμό. Πρακτικά τώρα. Οι υπηρεσίε express δεν περιορίζουν τον αριθμό των θεμάτων που μπορούν να μετακινηθούν από ένα αποστολέα σε έναν ε, παραλήπτη. πολλές φορές συζητώντας με διάφορες γενικές αρμόδιες διευθύνσεις, όταν μιλάτε για ένα μικρό φορτίο, ε, δύσκολα μπορούμε να ενταχθούμε. Δηλαδή από την άποψη της εταιρεία ε, προβήκαμε στη διανομή του iPad. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για μικρό φορτίο η διανομή του iPad. Συνεπώς, πρέπει να υπάρξει ένα σωστός ορισμός για το μικρό φορτίο και πρόσφατα πήγα σε μια επιτροπή που ασχολήθηκε με αυτό το θέμα, ίσως όχι στο ίδιο πλαίσιο, όπως για τα πνευματικά δικαιώματα, αλλά κατέληξαν ότι ο όρος πρέπει να τροποποιηθεί και να γίνει low value consignment, χαμηλής αξίας φορτίο. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με όλες τις υπηρεσίες της αρμόδιας και σας ευχαριστώ που μας δώσατε τη δυνατότητα να τοποθετηθούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ, σε ευχαριστώ Κίθ. Έχεις ε, πολύ σαφή τοποθέτηση. Ε, έθεσες πολλά σημαντικά ερωτήματα. Ξέχασα να πω ότι έχουμε εδώ μαζί μας και μια μεγάλη ομάδα από την Κομισιόν στελέχη τα οποία έχουν επεξεργαστεί σε βάθος το θέμα. Θα δώσω την ευκαιρία αργότερα στην Κομισιό να σχολιάσει. Ας προχωρήσουμε τώρα στον τελευταίο ομιλητή. Καλωσορίζω τον Κι Κοστέλο, που είναι αναπληρωτής διευθυντής ε, των Βρετανικών Τελωνίων. Ε, πολλοί συναδελφοί σας μας έχουν βοηθήσει ε, και θα ήθελα τώρα να σας δώσω το λόγο για να μας δώσετε τη δικιά σας τοποθέτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Κέβιν Κοστέλο. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία να απευθυνθώ στην Επιτροπή σας για τον αντίκτυπο στους ε, καταναλωτές των μικρών αυτών θεμάτων. Θα προσπαθήσω να καλύψω εν συντομία τους τομείς αυτούς. Καταρχάς, πολλά ακούσαμε ήδη για τα μικρά δέματα θα δείτε ότι το πρώτο σημείο που περιλαμβάνω στη διαφάνεια είναι ότι δεν υπάρχει ακόμα σωστός ορισμός για τα μικρά δέματα. Θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη για κάποιο είδους ε, ορισμό. Τι σημαίνει μικρό στην αξία, μικρό στο πάρο, στο, στις διαστάσεις. Ή ένα συνδυασμό στον Οσάνο. Θα θέλαμε να υπάρξει λοιπόν κάποιος ορισμός ε, για την νομοθεσία. Ακόμα και αν δεν είναι λεπτομερής, ο ορισμός αυτός θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για την επιλογή των κριτηρίων σε ό,τι αφορά την αξία, τον αριθμό των εμπορευμάτων, στο θέμα. Υπάρχουν διάφορα κριτήρια. Και ο κανονισμός δεν αναφέρεται καν στα κριτήρια της απόφασης αυτής. Το άλλο θέμα για τα μικρά δέματα. Η ανάγκη να εξισορροπηθούν τα δικαιώματα των επιχειρήσεων, των καταναλωτών, των οικονομικών ε, φορέων. Δεν είναι σαφές ε, ποια είναι η θέση για το παράλληλο εμπόριο σε ό,τι αφορά τα μικρά πακέτα, όπως και να οριστούν αυτά. Δεν θα θέλαμε να παρέμβουμε στο δικαίωμα του τελικού καταναλωτή να αγοράζει στη χαμηλότερη δυνατή τιμή ε, πρωτότυπα προϊόντα. Ξέρω ότι οι επιχειρήσεις προφανώς θα χρεώσουν ό,τι μπορούν και αυτό αποτελεί εμπορική πρακτική. Είναι ο ρόλος των ε, τελωνίων να υποστηρίξουν τις διαδικασίες αυτές μέσω συνοριακών ελέγχων για τέτοιες συμβατικές ε, σχέσεις. Θα πρέπει λοιπόν να εστιαστούμε στα παραποιημένα προϊόντα. Έχουμε κάποια στατιστικά στοιχεία. Μας έδωσε και κάποια στοιχεία ο συνάδελφος. Θα προχωρήσω, γιατί ουσιαστικά σε ό,τι αφορά τον όγκο των ε, υποθέσεων ταχυδρομικών δεμάτων και δεμάτων courier ε, μιλάμε για το μεγαλύτερο όγκο των περιπτώσεων παραβίασης, 51.000 περιπτώσεις, 64% όλων των περιπτώσεων παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, σε ό,τι αφορά το σύνολο των εμπορευμάτων, ε, μιλάμε για 5% των ε, παραποιημένων προϊόντων που εισάγονται, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, σε ό,τι αφορά την ε, απειλή για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις προέρχεται κυρίως από τις ε, μεγάλες αποστολές. Αν και είναι δυσανάλογος ο όγκος εργασίας που προκαλείται από τα μικρά δέματα. Βλέπουμε λοιπόν στα ταχυδρομικά δέματα ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα γιατί περιλαμβάνουν φαρμακευτικά προϊόντα, καλλιντικά, προϊόντα φροντίδας του σώματος, λοσιών, κρέμες και το καθεξής σε ό,τι αφορά τις αποσκευές των επιβατών. Βλέπουμε ότι εντοπίζουμε ετικέτες που προορίζονται για χρήση σε παραποιημένα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί η τελική διαδικασία ενδεχομένως να λαμβάνει χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα με την τοποθέτηση των ετικετών αυτών. Χρειάζεται λοιπόν έλεγχος κατά την εισαγωγή. Τώρα σε ό,τι αφορά τα μικρά δέματα, δεν αποτελούν όπως σας είπα μικρό πρόβλημα γιατί μπορεί να απορροφούν σημαντικούς πόρους των τελωνίων και επίσης ε, ανησυχούμε ιδιαίτερα για τις διαδικασίες που προσφέρονται και στους δικαιούχους, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχει υπερβολικό φόρτος, ε, υπερβολικός φόρτος και για τα τελωνία. γιατί ε, με τις διάφορες ε, προθεσμίες που δίδονται στους διάφορους φορείς είναι τεράστια η γραφειοκρατία, είναι τεράστια το γραφειοκρατικό άκτο και τεράστια κυχωρία αποθήκευση που γεμίζουν με τα εμπορεύματα αυτά. Και δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι πρόκειται σύντομα να υπάρξει μείωση στην ποσότητα, στον όγκο των διαδικτυακών πωλήσεων. Άρα σίγουρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Προβλήματα. Η πολύ ψηλό όγκο ε, δεμάτων χαμηλή αξία. Αλλά χαμηλής αξίας και σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους και σε ό,τι αφορά την προσπάθεια που διατίθεται, προτίθεται να καταβάλουν. Όταν ο παραλήπτης ε, καταγγέλει την κατάσχεση και δηλώνει ότι δεν είναι παραποιημένα τα προϊόντα, συνήθως πάντα οι δικαιούχοι δεν λαμβάνουν μέτρα γιατί ακριβώς είναι τόσο χαμηλή η αξία των εμπορευμάτων. Άρα Οπότε δεν υπάρχει αμφισβήτηση της κατάσκησης. Ε, προβαίνουμε σχεδόν πάντα σε καταστροφή των εμπορευμάτων και όποτε γίνεται τέτοια αμφισβήτηση, ε, με σχεδόν πάντα διατίθενται στην αγορά τα προϊόντα αυτά. Πρόκειται για ένα δίκτυο, ένα κύκλο κλίματα εγκλήματος, να μην το ξεχνάμε αυτό. Το να πολύ κανείς ε, ε, εμπορεύματα από το εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ πιο εύκολο από ότι το να έχει έδρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουμε υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί πρωτεύοντα στόχο. Θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία λοιπόν μεταξύ των αναγκών των πολιτών, των επιχειρήσεων. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα παραποιημένα προϊόντα είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία, προβλέπει μια ιδιαίτερη διαδικασία που θα καταστήσει πιο εύκολη την ε, ε, διαδικασία που ακολουθούν τα τελωνία. Ο δικαιούχο, όπω είπαν οι συνάδελφοι, θα πρέπει να αποφασίζει κατά πόσο πρόκειται ή όχι για παραποιημένα προϊόντα και αν θέλει να κάνει αίτηση για να συμπεριληφθούν και τα ιδιωτικά μικρά πακέτα, θα πρέπει να είναι σαφής για το πώς θα λαμβάνουν τις αποφάσεις τους στην τελωνία. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, τα πράγματα είναι απλά, γιατί ο δικαιούχος μας λέει, για παράδειγμα, ότι δεν κατασκευάζουμε στην Κίνα, οτιδήποτε έρχεται από Κίνα είναι παραποιημένο. Αλλά σε πολλές ε, περιπτώσεις ε, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, γιατί πολλά γνήσια προϊόντα κατασκευάζονται στην Κίνα. Αναφέρθηκα στο δικαίωμα του να εισακούεται κανείς. Μας ανησυχεί ο αντίκτυπος στο δικαίωμα αυτό, είτε πριν είτε μετά την ανάληψη δράσης. Και ανησυχούμε σε ό,τι αφορά την ε, ε, επιφόρτηση σε ό,τι αφορά την ανάληψη του κόστους. Αυτό μπορεί να πέσει στους ώμους των πελωνίων σε ό,τι αφορά την ε, εξέταση και την καταστροφή των προϊόντων. Σε ό,τι αφορά ε, θέματα ενημέρωσης και θέματα πληροφόρησης, οι δικαιούχοι χρειάζονται πληροφορίες και όταν καταστρέφουμε μικρά δέματα, με απλοποιημένη διαδικασία. Είναι σημαντικό να έχουμε την ευελιξία να παρέχουμε τέτοιες πληροφορίες στους δικαιούχους προκειμένου να γνωρίζουν την έκταση του προβλήματος ακόμη και αν δεν είναι διδεθμένοι να λαμβάνουν σε κάθε περίπτωση ε, δράση και να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Αλλά τουλάχιστον θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για να προστατεύσουν περαιτέρω την, ε, τα προϊόντα τους. Σε ό,τι αφορά τέλος ε, τις αποσκευές των επιβατών των ταξιδιωτών. Μας ε, ανησυχεί η κατάσχεση μικρών ποσοτήτων παραποιημένων ε, προϊόντων. Το ότι κάποιος ε, ταξιδεύει στο εξωτερικό σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια έξοδα. Δεν θεωρούμε λοιπόν ότι είναι τόσο μεγάλο ο κίνδυνο σε σχέση με άλλες μορφές εισαγωγών. Καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να καταπολεμηθούν οι εμπορικέ εισαγωγέ, σε ό,τι αφορά τι αποσκευέ, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τα κοσμήματα, σε ό,τι αφορά προϊόντα παραποιημένα και ε, παραποιημένες ετικέτες. Και σκοπό θα πρέπει να είναι η καταπολέμηση των ε, δραστηριοτήτων εισαγωγή παραποιημένων προτεραιοτήτων με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κλείσω λοιπόν στο σημείο αυτό. Ξεπέρασα ελαφρώς τα 10 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Μόλις ε, λίγα τεσσερά λεπτά. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας και πολλοί εξημών δεν είχαν σκεφτεί ότι μπορούν ε, οι επιβάτες στις αποσκευές τους να μεταφέρουν πλαστές ετικέτες. Είχα υποσχεθεί στον κύριο Τεκάμπος να πάρει πρώτα στο λόγο και είχα, ε, αν θέλει φυσικά και ο εισηγητής να πάρει στο λόγο, ε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εγώ καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω το συνάδελφο που, που διοργάνωσε αυτή την ακρόαση και μας έδωσε την ευκαιρία να ακούσουμε αυτούς τους εξαίρετους ομιλητές που μπαίνουν στην ουσία του θέματος. Οι δικές μου ανησυχίες εν μέρη ε, καλύφθηκαν από το τελευταίο τελευταίο γύρο παρεμβάσεων που θεωρεί πως ένα από τα κεντρικά προβλήματα είναι ο ορισμός του μικρού δέματος. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι αναπόφευκτο. Πρέπει να εμβαθύνουμε στην έννοια αυτή. Αλλά σε σχέση με την καταστροφή το δικαίωμα καταστροφής ε, των μικρών δεμάτων, εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε να δούμε αν θέλουμε να ακολουθήσουμε μια αναλυσίδα που είναι ταυτόχρονα αρκετά μεγάλη αλλά και αρκετά μικρή. Δηλαδή, είναι μεγάλο το δίχτυ για τα, φαρμακευτικά προϊόντα, αλλά στενό για όλα όσα αφορούν το, το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και όταν λέω ηλεκτρονικό εμπόριο δεν σημαίνει ότι το καταδικάζω, όχι, γιατί το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει να κάνει με ανταλλαγή υπηρεσιών ή αγαθών εντός της Ένωσης, αλλά μπορεί να υπάρχει και εμπόριο ηλεκτρονικό με προϊόντα εισαγόμενα και μπορεί να υπάρχουν ε, εισαγωγής, ε, διαμεσολάβηση, άμεση παράδοση, άμεση παράδοση μικρών δεμάτων στον καταναλωτή εντός της Ένωσης. Άρα λοιπόν ε, μπλεκόμαστε και εδώ ξέρω πως θα υπάρξει και τρίτος γύρος της συζήτηση για τα φάρμακα γενικής ε, ονομασίας. Εγώ δεν θα μπορέσω να παρακολουθήσω το θέμα αυτό, αλλά ίσως είναι και το πιο καυτό και το πιο δύσκολο. Επίσης, ε, έχω μια περιέργεια να γνωρίζω στη Γερμανία αυτή η ξαφνική αύξηση γιατί υπήρξε μια τρομερή εχμή το 2010 ε, για τις κατασχέσεις, τι είδους προϊόντα αφορά. Είπατε ότι είναι, είναι φάρμακα. Θα μου πείτε. Ε, συνοψίζοντας, έχουμε να κάνουμε μια νομοθεσία που πρέπει να αντιμετωπίσει διάφορα παράδοξα σχήματα, διότι, όπως είπα, η αλυσίδα είναι, ο κρίκος μάλλον σε αλυσίδα θέλουμε να είναι πολύ στενός, αλλά αν είναι πολύ στενός, πολύ μικρό, θα βλάψουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο. Θέλουμε ε, επίσης ο κρίκος αυτός να είναι, αν μάλλον αυτός ο κρίκος είναι πολύ ευρύς, πολύ φαρδής, δεν θα καλύπτει κάποια προϊόντα τα οποία μπορεί να είναι βλαβερά για την υγεία, όπω τα φαρμακευτικά. Ωστόσο πιστεύω πω η δουλειά αυτή θα εξελιχθεί, θα εξελιχθεί με βάση τα άρθρα 24 και τα συναφή που έχει να κάνει με τις παραγγελίες μικρής αξίας, τον καθορισμό όλων αυτών των ενιών, γιατί διαφορετικά μπορεί να έχουμε παρενέργειες μιας ε, τέτοιας νομοθεσίας, την οποία κατά άλλα όλοι μας θέλουμε να υποστηρίξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χέντ που είναι σκιώδης εισηγήτρια για την πρόταση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω διερμηνία από τα Σουηδικα, προς τα Σουηδικά, αλλά μου είπαν ότι μπορώ να μιλήσω Σουηδικά. Φωνάξτε μου αν <laughs> μπορείτε να με καταλάβετε η πρόπτικη του καταναλωτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για μένα. Σήμερα το πρωί συζητήσαμε ειδικότερα τους ευάλωτους καταναλωτές. Είναι πολύ σημαντική μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Δεν πρέπει να τους ξεχνούμε. Μιλάμε για τα παιδιά, μιλάμε για τους ασθενείς και για προϊόντα όπως τα παιχνίδια, τα φαρμακευτικά, τα τρόφιμα. Μπορεί πραγματικά να είναι επικίνδυνα για τους ανθρώπους, τους ευάλωτους. Είχα την ευκαιρία να πάω στη Σανγκάη το 2008 και επισκέφθηκα τους τελωνιακούς εκεί και ο πρόεδρος ήταν μαζί σε αυτή την αποστολή και πρέπει να πω ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα πράγματα. Πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με τρίτες χώρες για να σταματήσουμε αυτά τα προϊόντα να εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα αντιμετωπίσουμε τα, τις ε, χώρες καταγωγής. Πρέπει να σταματήσουμε την παραγωγή αυτών των προϊόντων και την, να αποτύχουμε την καταστροφή. Η πραγματική μου ερώτηση απευθύνεται στην Κομισιό. Αν βέβαια κάποιος άλλος έχει απάντηση, ακόμη καλύτερα. Αφορά τους ορισμούς. Δεν έχουμε ορισμούς. Δίνω ένα παράδειγμα. Τι εννοούμε με προϊόντα που μπορεί εύκολα να καταστραφούν. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα τι σημαίνει ένα μικρό φορτίο, η δέμα. Η Κομισιόν δεν έχει προτείνει ορισμούς γι' αυτά. Αυτό που λέει είναι ότι θα υπάρξει πράξη εξουσιοδότησης, αλλά δεν είναι καλύτερο να έχουμε έναν ορισμό στην οδηγία. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Έντουιν θα ήταν ο τελευταίος ομιλητής μας. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θα θέλουν το λόγο. Όχι. Λοιπόν, σχολιάσουν οι συμμετέχοντες στο πάνελ. Αρχίζουμε με τον κύριο Κοστέλο. Δώστε μας τα σχόλιά σας. Κύριε Κοστέλο, πρώτος. Πάνω όσα έλεγχτε. Σύμφωνο με την προηγούμενη ομιλήτρια. Οι ενέργειες των τελωνίων των Βρετανικών δίνουν προτεραιότητα στα προϊόντα τα οποία μπορούν να βλάψουν τους ανθρώπους. Ακόμη πολλά εξαρτώνται και από τους άλλους υφιστάμενους κινδύνους. Αυτή τη στιγμή τα προϊόντα, τα παραποιημένα, τα, ο μεγαλύτερος όγκος είναι τα τσιγάρα τα οποία ε, προέρχονται από την Κίνα κατάσχονται ε, λόγω φόρου κατανάλωσης. Ε, Βεβαίω, επειδή διώκουμε συνεχώς αυτό το εμπόριο, γι' αυτό βρίσκουμε και τόσα παραποιημένα. Καμιά φορά ανοίγουμε για να βρούμε καπνό και βρίσκουμε φουστάνια και βεβαίω δεν μπορούμε να τα ξανακλείσουμε και να τα στείλουμε, να τα αφήσουμε να φύγουν. Πρέπει να ενεργήσουμε. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, αν δεν είχαμε πρόβλημα με τον κινέζικο καπνό, τότε δεν θα βρίσκαμε και τόσες απομιμήσεις. Η έλεγχη στα σύνορα, ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με μικρά φορτία και πακέτα, η έλεγχη στα σύνορα θα είναι πάντα ένας μη αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος. Πρέπει να συνεργαστούμε με τις κινέζικες αρχές και διάφορες δικαιοδοσίες για να σταματήσει το πρόβλημα εκεί. Πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε στο διαδίκτυο να μην διαφημίζονται αυτά τα προϊόντα και πρέπει να επιμορφώσουμε και τους καταναλωτές. Έχουμε ένα πρόγραμμα δράσης με την Κίνα για να προχωρήσουμε και ε, έχουν υλοποιηθεί διάφορες ενέργειες. Δεν, ο έλεγχος στα σύνορα δεν τα καλύπτει όλα. Ο, κύριο, ο κύριος Όλ τώρα. Δεν έχω πολλά σχόλια. Ο καθηγητής Κάμπος αναφέρθηκε σε ένα ε, δίχτυ στενά ανοίγματα. Αυτό με ανησυχεί. Ε, τα τελωνία θα πρέπει να είναι η τελευταία λύση για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Στα 27 κράτη-μέλη ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα είναι το εξής. Δεν έχουν τα τελωνία τους πόρους για να αντιμετωπίσουν το μέγεθος του προβλήματος. Από την επιχειρηματική πλευρά κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά βεβαίως δεν μπορούμε να ανοιχνεύσουμε τα παραποιημένα, απαραίτητο και τις απομιμήσεις, αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι, αν μας λεχθεί ότι ένας αποστολέας στέλνει τέτοια φορτία, μπορούμε να τα σταματήσουμε και να κλείσουμε το λογαριασμό του. Διότι το τελευταίο που θέλουμε, θέλουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι να τους κλείσει το λογαριασμό τους, την επιχείρησή του. Υπάρχει μεγάλος αριθμός φορτίων που δεσμεύονται στις αποθήκες μας και μόλις έχουμε τους πόρους να αντιμετωπίσουμε το θέμα και να προχωρήσουμε, θα πετύχουμε. Όταν θα μπορέσουμε δηλαδή να συνεργαστούμε πραγματικά με τις χώρες καταγωγής. Αυτό θα είναι το πιο αποτελεσματικό. Έχει τεράστια εμπειρία και το θέμα των τελωνιακών πόρων βεβαίως δεν είναι κάτι που μπορούμε να ρυθμίσουμε. Είναι θέμα των κρατών μελών. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει συνεχής, μια συνεχής πίεση για αύξηση ανθρωπίνων πόρων και άλλων πόρων. Κατάλαβα από όλες αυτές τις παρεμβάσεις ότι υπάρχει πρόβλημα ενιών, μικρά δέματα, μικρά φορτία κτλ. Όταν απαντήσαμε στην περίοδο συνδιαλλαγής για αυτό το νομοθέτημα, προσπαθήσαμε να βρούμε, βρούμε κάποιους προσανατολισμούς και να εμπνευστούμε, μια και ασχολούμεθα με το ταχυδρομείο, από τους ορισμούς της Παγκόσμιας Ένωσης Ταχυδρομείων. Εκεί υπάρχει ορισμός για το τι είναι μια επιστολή, τι είναι ένα μικρό δέμα, ε, πώς έχει συσκευαστεί, τι βάρος έχει λοιπά. Λοιπόν, δεν λέω ότι μπορούμε αυτά να τα μεταφέρουμε στο δίκαιό μας άμεσα. Όμως, το μέγεθος και το βάρος είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε ένα εμπορευματοκιβώτιο και τα διάφορα μικροδέματα για αποστολή εξπρές κατευθυντήριες γραμμές λοιπόν θα μπορούσαν να εμπνευστούν από όσα έχει εφαρμόσει η Παγκόσμια Ένωση Τοχυδρομείων. Τώρα, να καταστρέφονται εύκολα. Τι θα πει αυτό, με χαμηλό κόστος φαντάζομαι. Μιλήσαμε για τον καπνό και την παραποίησή του. Ξέρουμε ποιο είναι το οικολογικό κόστος της καταστροφής του καπνού, είναι επικίνδυνο και δεν το καταστρέφουμε όπως ε, να είναι, πρέπει να το ποτίζουμε τακτικά για να μην ανάψει πυρκαγιά κτλ. Το ίδιο ισχύει για το ενόπνευμα. Ε, χρειαζόμαστε συγκεκριμένη επεξεργασία για να πετύχουμε την καταστροφή. Χρειάζεται δηλαδή και εξοπλισμός. Είναι σαφές συνεπώς ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην καταστροφή κάποιων δεμάτων και την καταστροφή μιας μάζας ολόκληρης κάτω από οικολογικές συνθήκες. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους τελωνιακούς και τους δικαιούχους. Ε, ε, μπορούν να βρεθούν ε, βεβαίω ενδιαφέρουσε λύσεις. Τώρα, όσον αφορά τις κατασχέσεις, ενδύματα και ηλεκτρονικά και τσιγάρα. Αυτέ είναι οι βασικές κατασχέσεις μας. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα περνάμε στην τελευταία συνεδρία. Α, ο κύριος Τόλαρ, με συγχωρείτε. Σας ευχαριστώ. Ήθελα να απαντήσω στην άμεση ερώτηση του Γερμανού συναδέλφου, μάλλον για τη Γερμανία. Ποιες αποστολές προκάλεσαν αυτή τη τεράστια αύξηση και αν πρόκειται μόνο για ε, φάρμακα. Όχι, δεν πρόκειται μόνο για φάρμακα. Βλέπουμε σε περίπου 540 περιπτώσεις αποστολές φαρμάκων μέσω ταχυδρομείου. Πρόκειται για φάρμακα για επιδόσεις τις οποίες ε, συνειδητά ο καταναλωτής τα αγοράζει μέσω του διαδικτύου γνωρίζοντας ότι δεν πρόκειται για νόμιμα προϊόντα και διαπιστώνουμε επανειλημμένα ότι η διαφορά της τιμής ε, οδηγεί τον καταναλωτή να δέχεται τα ενδεχόμενα, τις ενδεχόμενες επιπτώσεις για την υγεία του. Η αύξηση το 2010 είχε να κάνει με το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η Ταϊλάνδη έκανε και μεγάλα βήματα προς τα εμπρός και φαίνεται ότι πολύ συχνά οι καταναλωτές θεωρούσαν ότι ήταν πολύ ακριβό ε, ένα ενθύμιο, 80 ευρώ, και γι' αυτό λοιπόν προτίμησαν τα παραποιημένα. Right. Well, thank you very much indeed for that deceptively simple explanation. <laughs> Σας ευχαριστώ για την απλή αυτή εξήγηση. Θα έχουμε και τους Ολυμπιακούς ε, φέτος θα έχετε πολλά να κάνετε. Νομίζω ότι πάντα υπάρχουν διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις ε, που θα αποτελούν αφορμή για τέτοιες ε, δραστηριότητες. Τώρα, θα κοιτάξουμε άλλο ένα θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα εμπορεύματα σε διαμετακόμιση. Τέσσερις ομιλητές. Αν θα μπορούσα να σας παρακαλέσω να τηρήσετε τα χρονικά όρια. Δυστυχώς, ο Γενικός ε, διευθυντή ε, τη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Προϊόντων δεν μπορέσει να παραβρεθεί, αλλά ο Χιου Πούλεν, ο οποίο είναι αρμόδιο για θέματα εξωτερικού εμπορίου του Λουξεμβούργου, θα τον αντικαταστήσει. Και μοναδικό όρο που του θέτει είναι να μην μιλήσει παραπάνω από 10 λεπτά. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κάθε προσπάθεια να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Ρίτσαρτ Μπέκστραμ, ο οποίος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Είμαι αντιπρόεδρος της ομάδας εργασίας κατά των παραποιημένων προϊόντων. Έχω λοιπόν κάποια εμπειρία για τα θέματα αυτά. Δύο λόγια. Καταρχάς, για την Ομοσπονδία μας που εκπροσωπεί την καινοτόμα φαρμακευτική βιομηχανία της Ευρώπης 31 εθνικές ενώσεις ε, φαρμακοβιομηχανίας εκπροσωπούμε και εκπροσωπούμε 600.000 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη περίπου. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τα προϊόντα σε διαμετακόμιση και να κάνουμε κάποια σχόλια και για τα άλλα θέματα που ε, ακούσαμε. Η Ομοσπονδία μας ε, καταπολεμά εκτεταμένα τέτοια προϊόντα και βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, παραπημένα φάρμακα τα οποία περιλαμβάνουν τεστ, δεν έχουν δραστικές ουσίες. Τα βλέπουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε άλλα μέρη στον κόσμο και αποτελούν πολύ σημαντική απειλή στην υγεία των ασθενών. Συνεπάγονται και θανάτους πολλές φορές των ασθενών. Νομίζω ότι η απειλή των παραποιημένων σε ό,τι αφορά τα προϊόντα στη μετακόμιση είναι ιδιαίτερα μεγάλη και η Παγκόσμια Οργάνωση υπολογίζει υγείας υπολογίζει ότι το 1 τρίτο των φαρμάκων στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι παραποιημένα. Είναι σαφές ότι η μεγάλη πλειοψηφία, πλειονότητα των ε, εμπορευμάτων αυτών, των φαρμάκων αυτών δεν ε, παρασκευάζονται επί τόπου, μεταφέρονται από άλλες χώρες και βλέπουμε ότι η Ευρώπη χάρη στην ε, γεωγραφική της θέση έχει καταστεί κόμβος για τη μεταφορά των εμπορευμάτων αυτών και έχουμε δει παραδείγματα όπου στο αεροδρόμιο των ε, Βρυξελών έγινε κατάσχεση ε, φαρμάκων κατά της Ελληνοσίας που δεν περιλαμβάνουν δραστικές ουσίες. Αυτό είναι κρίσιμη σημασία γιατί σημαίνει ότι ο κόσμος που τα λαμβάνει τα φάρμακα αυτά δεν ακολουθεί τελικά θεραπεία και αυτό ασφαλώς πολύ εύκολα μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο των ασθενών αυτών αλλά υπάρχει και γενικότερη ανησυχία ότι θα υπάρχει αυξανόμενη αντίσταση στα φάρμακα κατά της ελονοσίας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα αντιβιωτικά. Άρα, νομίζω ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να τις αναλάβουμε στα σοβαρά σε ό,τι αφορά την μεταφορά μέσω Ευρώπης τέτοιων φαρμάκων. Και με ιδιαίτερη ανησυχία είδαμε το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο δεν περιλαμβάνει ουσιαστικά αναφορά ρητή στην ε, ανάγκη ε, διεξαγωγής ελέγχου σε τέτοια εμπορεύματα στην Ευρώπη. Θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα θέμα δημόσιας υγείας, κρίσιμο μάλιστα και κατά συνέπεια είναι πάρα πολύ σημαντικό τα εμπορεύματα να υπόκεινται στους σωστούς ελέγχους. Αυτό το θέμα θα έπρεπε να είναι ουσιαστικά μη αμφιλεγόμενο, αλλά δυστυχώς λόγω διαφόρων περιστατικών που σημειώθηκα το 2008 με την ε, κράτηση διαφόρων προϊόντων που παραβίαζαν διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Ε, το θέμα αυτό έχει καταστεί αμφιλεγόμενο. Θα ήθελα να πω ότι η Ομοσπονδία μας δεν έχουν οποιαδήποτε συμφέρον και δεν θέλουν να ε, σταματήσουν την εμπορία νόμιμων νόσιμων φαρμάκων. Δεν μας αφορά καθόλου αυτό. Ε, προβήκαμε μάλιστα προβήκαμε σε μια σχετική δήλωση το 2009 η οποία διασ... έκανε σαφή την ε, θέση μας. Θεωρούσαμε λοιπόν ότι περιοριζόμαστε, περιορίστηκε μάλλον το περιστατικό αυτό σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις, αρχές του 2009, τέλη του 2008, ανησυχούμε για καθυστερήσεις που προκλήθηκαν λόγω των ελέγχων ε, που επιβλήθηκαν. Σε περίπτωση όμως ε, που δεν υπήρχε λόγος να εμποδιστεί η μεταφορά των προϊόντων, ε, απελευθερώθηκαν για διάθεση στην αγορά. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι και όπου είναι απαραίτητο να γίνεται κατάσχεση και καταστροφή των ε, προϊόντων αυτών. Δεν ε, ε, θέλουμε όμως να σταματήσουμε την εμπορία νόμιμων γεννόσιμων φαρμάκων. Τώρα, μερικά σχόλια για τα άλλα θέματα που ακούσαμε σήμερα το απόγευμα, για τα μικρά δέματα. Προφανώς, είναι προς το συμφέρον το δικό μας να διευκρινιστεί ο όρος, γιατί τα φάρμακα είναι και ελαφριά και μικρά σαν διαστάσεις και μπορεί να έχουν υψηλή αξία. Όπως είπαν διάφοροι ομιλητές, ο μεγάλος όγκος τέτοιων ε, αποστολών και τέτοιων δεμάτων έχει να κάνει με την διάδοση των ε, φαρμακείων στο διαδίκτυο. 68% των ε, δεμάτων παραποιημένων εμπορευμάτων αποτελούν τα φάρμακα. Αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα εκατομμύριο τέτοια εμπορεύματα κατασχέθηκαν σε τρεις ημέρες. Αυτό νομίζω ότι καταδεικνύει την κλίμακα του προβλήματος. Και έχοντας επισκεφτεί το αεροδρόμιο της ε, Φραγκφούρτης, μου ανακοίνωσαν οι τελωνιακοί ότι ε, έκαναν κατάσχεση 30 έως 50 φακέλους κάθε μέρα με παραποιημένα φάρμακα. Νομίζω ότι η κλίμακα μιλάει από μόνη της και υποστηρίζουμε λοιπόν την εισαγωγή μιας τέτοια διαδικασίας που θεωρούμε ότι θα καταστήσει πολύ πιο απλή και σαφή τη διαδικασία κατάσχεσης και καταστροφής των προϊόντων αυτών. Νομίζω και πάλι ότι οι απειλές για την υγεία δεν μπορούν να παραμεριστούν. Ε, πρέπει να τις λάβουμε σοβαρά υπόψη. Μας είπαν ότι για κάθε φάκελο που κατάσχουν μπορεί να χρειάζεται και 45 λεπτά ε, χαρτοδουλιά μετά. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο όγκος. Κάτι άλλο τώρα για την ανταλλαγή πληροφοριών. Πολλοί ομιλητέ μίλησαν για την ανάγκη να εξεταστεί και να αντιμετωπιστεί η πηγή του προβλήματος. Και σε ό,τι αφορά τις ε, αποστολές, τις εισερχόμενες. Είναι σημαντικό τα τελωνία να μοιράζονται όσο πιο πολλές πληροφορίες γίνεται για τους εγκληματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό προκειμένου να κλείσουν τα φαρμακεία αυτά στο διαδίκτυο. Μία σχετική μελέτη πρόσφατα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 62% των φαρμάκων που αγοράζονται από παράνομα διαδικτυακά φάρμακα ήταν παραποιημένα. 95% των φαρμακείων αυτών δρούν παράνομα. Άρα υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη συνεργασίας για να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε η ανάγκη συνεργασίας και με τους ε, ενδιάμεσους φορείς σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, προκειμένου να συνεργαστούμε για να σταματήσουν οι αποστολές αυτές, τα δέματα αυτά, να σταματήσουν οι υπηρεσίες παροχής πληρωμών, μεταφορών σε αυτά τα φαρμακεία. Θεωρώ λοιπόν ότι η ανταλλαγή πληροφοριών είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο το οποίο θα πρέπει να καλύπτεται και θα ήθελα τώρα στο σημείο αυτό να κλείσω επαναλαμβάνοντας το εξής. Τα εμπορεύματα σε διαμετακόμιση αποτελεί σημαντικό, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό τομέα που λείπει από την νομοθεσία ο ρόλος και η ευθύνη της Ευρώπης για την πρόληψη ε, του κινδύνου αυτού της υγείας ε, θα πρέπει να αναγνωριστεί. Γιατί φαίνεται ότι μπορούμε να πάρουμε πολλά βήματα για να προστατεύσουμε την υγεία των Ευρωπαίων ασθενών, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να λάβουμε τα παρόμοια μέτρα για να προστατεύσουμε τους ασθενείς σε παγκόσμιο επίπεδο. Θεωρούμε κατά δεύτερον ότι τα μικρά δέματα αποτελούν ένα κρίσιμο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε την πλημμυρίδα παράνομων φαρμάκων που εισέρχονται στην Ευρώπη και θα πρέπει να καταπολεμηθούν τα παράνομα φαρμακεία online και τέλος ανταλλαγή πληροφοριών η οποία θα επιτρέψει, θα επιτρέψει σε όλους τους ε, μεσάζοντες να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να καταπολεμήσουν την απειλή. Θα ήθελα λοιπόν πρόεδρος στο σημείο αυτό να κλείσω και να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακριβώς την ώρα σας. Μας δώσατε τροφή για σκέψη. Να μείνουμε στην φαρμακοβιομηχανία με την επόμενη ομιλήτριά μας που είναι η κυρία Λίβια Μάλο, κυβερνητική διευθύντρια στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ε, φαρμάκων γενικευμένου σήματος. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και που μου δίνετε την ευκαιρία να σας αναφέρω την άποψη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Είμαστε ε, έχει πάνω από χίλιες εταιρείε σε 34 ευρωπαϊκές χώρες. Ε, έχουμε υπολογίσει ότι μπορούμε να ε, παράγουμε 30 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στα κράτη-μέλη μας. Επίσης έχουμε υπολογίσει ότι απασχολούμε 150.000 ανθρώπους. Είμαστε ένας από τους πιο ανταγωνιστικούς τομείς αυτή τη στιγμή στην Ένωση και όταν ε, εκπνεύσει η ισχύουσα νομοθεσία τότε οι τιμές μπορεί να κατέβουν 30 με 90% όταν δηλαδή εκπνεύσει το δικαίωμα ευρεσιτεχνία. Ε, σας δώσουμε την άποψή μα για τον νέο κανονισμό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις ε, διάφορες υποθέσεις που συνέβησαν πριν από κάποια χρόνια. Καταρχήν, η παγκοσμιοποίηση της παραχάραξης και πωλήσει μέσω ίντερνετ, πολύ σημαντικές νέες προκλήσεις και προβλήματα. Να γνωρίζουμε ε, το σημαντικό ρόλο των τελωνιακών αρχών στα κράτη-μέλη και επίσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ώστε να αναχαιτήσουν ε, την εισαγωγή παραχαραγμένων προϊόντων για να προστατεύσουν την υγεία των καταναλωτών. Η παραχάραξη, η παραποίηση φαρμάκων είναι εγκληματική πράξη που θέτει σε κίνδυνο την ζωή των ασθενών. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να προστατευτούν οι καταναλωτέ από αυτά. Αντίθετα με τα παραχαραγμένα ή τα παραποιημένα φάρμακα, τα, τα, τα φάρμακα γενικευμένης ε, σήμασης ε, πρέπει να είναι τόσο καλά όσο και τα αυθεντικά. Αντίθετα, τα παραποιημένα είναι κατώτερα ε, πλαστά προϊόντα που δεν πληρούν καμία προδιαγραφή και αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Επανέρχομαι στο θέμα της παραποίησης. Λόγω αυτού του ευρύτατου θέματος παραποίησης, τα θεμητά, τα καλή πίστης ε, ε, σήματα, συγγνώμη, φάρμακα με γενικευμένο σήμα έχουν ε, ε, κακώς παρακρατηθεί. Να σας δώσω μια περίπτωση πολύ γνωστή που έγινε στην Ολλανδία. Τι συνέβη. Υπήρξαν ε, διάφορα φορτία τα οποία κατασχέθηκαν από διάφορες εταιρείες που πήγαιναν στη Βραζιλία, την Κολομβία και το Περού. Αυτό που συνέβη ήταν το εξή. Το δικαστήριο στις κάτω χώρες θεώρησε πως ε, ήταν ότι είχαν παραβιάσει την ευρεσιτεχνία επειδή υποτίθεται ότι είχαν κατασκευαστεί στην Ολλανδία που ίσχυε ακόμα η ευρεσιτεχνία. Ο τύπος απλώς είπε ότι πρόκειται για παραποιημένα φάρμακα και αυτό έδωσε μια πολύ άσχημη εικόνα στη βιομηχανία των ε, φαρμάκων γενικευμένου σήματος. Όπως ξέρετε αυτό προκάλεσε ε, επεισόδιο μεταξύ της Ένωσης και της Βραζιλίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να αντιμετωπίσει το θέμα προτείνοντας νέο κανονισμό. Και θα σας πω ποιες είναι οι απόψεις μας περί αυτού. Επόμενη διαφάνεια. Το θέμα της διάλευσης ε, αντιμετωπίζεται στο προήμιο στην παράγραφο 17 στη νέα πρόταση. Εμείς αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι τα τελωνία όταν εκτιμούν μια πιθανή παραβίαση ενός δικαιώματος πνευματικής διοκτησίας θα σταματήσουν τα φάρμακα μόνο αν υπάρχει ουσιαστική πιθανότητα τα αγαθά αυτά να ξαναμπούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Το πρόβλημα αυτό αφορά μόνο τα φάρμακα. Εμείς το στηρίζουμε αυτό, αλλά πιστεύουμε πως δεν είναι αρκετά ξεκάθαρο. Φοβούμαστε ότι τα τελωνία δεν θα είναι σε θέση να καθορίσουν αν όντω υπάρχει πιθανότητα ε, εισόδου τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε περισσότερες κατευθυντήριες γραμμές, οδηγίες. Πώς θα γίνει κάτι τέτοιο μέσω κατευθυντηρίων γραμμών, μέσω κάποιου άρθρου. Ε, το πρέπει να το συζητήσει το Κοινοβούλιο. Εμείς προτείνουμε ως κλάδος, την επόμενη διαφάνεια παρακαλώ, αυτέ, αυτές οι οδηγίες να ξεκινούν ως εξή. Ότι δηλαδή τα τελωνία θα πρέπει να είναι σε θέση να έρθουν σε επαφή με τον παραλήπτη και να επαληθεύσουν αν τα φάρμακα που θα παρακρατηθούν, θα κατασχεθούν, έχουν άδεια ε, ή αν είναι σε κάποιο κατάλογο υποκατάστατων. Αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, σημαίνει κανονικά πως το φάρμακο αυτό δεν θα κυκλοφορήσει στο συγκεκριμένο κράτος. Δεν θα πρέπει, να υπάρχει φόβος ότι αυτό θα φύγει, θα ε, ξαναμπεί στην αγορά. Επίσης, θέλαμε να προτείνουμε ο τελενιακός να ρωτήσει να ζητήσει από την ε, κατασκευάστρια εταιρεία μια επιστολή που να λέει πού κατευθύνεται το συγκεκριμένο φορτίο. Νομίζω πως έτσι θα μπορούσαμε να βοηθηθούν τα τελωνία. Ένα άλλο σημείο του κανονισμού είναι ο ορισμός. Εμείς εκτιμούμε ιδιαίτερα τις διαφορές που έχουν γίνει εδώ και τις διακρίσεις ανάμεσα στην παραβίαση ευρεσιτεχνία ή την παραποίηση του ίδιου του φαρμάκου. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες, ε, παραβίαση ευρεσιτεχνίας, πειρατεία, ε, παραποίηση ή παράνομη χρήση εμπορικού σήματος και υπάρχει και εκείνη η κατηγορία όπου εμείς εντασσόμαστε ως κατασκευαστές γενικευμένων ε, φαρμάκων Όταν δηλαδή υπάρχει υποψία παραβίασης ενός δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, δηλαδή κάποιας ευρεσιτεχνίας. Παραβίαση δηλαδή το πνεύματος ε, το, της ευρεσιτεχνίας δεν είναι ε, το ίδιο. Το να εξηγήσουμε τη διαφορά. Μια πλαστή τσάντα ή όλοι ξέρουμε πως είναι παραβίαση εμπορικού σήματος ο, όμως με τα φάρμακα δεν είναι το ίδιο ο δικαστής πρέπει να αποφασίσει μπορεί να, να περάσουν και τρία χρόνια μπορεί να κερδίσει την υπόθεση στη Βρετανία να τη χάσει στη Γερμανία και ούτω καθεξής είναι πολύ σημαντικό οι παραβιάσεις ε, της, ε, των ευρεσιτεχνών να μην θεωρηθούν εγκλήματα στον ίδιο βαθμό όπως η παραποίηση των φαρμάκων. Τώρα, το θέμα του εμπορικού σήματος ενός ιατρικού προϊόντος είναι παράνομο, μπορεί να είναι κίνδυνο κάτι τέτοιο για την ανθρώπινη υγεία. Επίσης υπάρχει, δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχει ρυθμιστική αρχή, ούτε ποιοτικό έλεγχος του προϊόντος και είναι μέγας ο κίνδυνος για τον καταναλωτή γιατί το, το φάρμακο μπορεί να σκοτώσει, μπορεί να μην περιέχει κάποιο ενεργό συστατικό και ούτω καθεξής. Έπειτα έχουμε την παραβίαση του, της ευρεσιτεχνίας συμβαίνει διαρκώς όσον αφορά την νόμιμη αλυσίδα παραγωγής και παροχής. Εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί τα φάρμακά μας είναι ε, αξιολογημένα και περνάμε και από διαδικασία ποιότητας. Υπάρχει δηλαδή διαφάνεια, θεμητός ανταγωνισμός και αυτό που βλέπουμε εδώ είναι μόνο μια εμπορική διαφορά όπου κάποιες φορές μπορεί να αμφισβητήσουμε μια ευρεσιτεχνία γιατί πιστεύουμε πως είναι άκυρη ή αδύναμη. Για να είναι ξεκάθαρα λοιπόν τα πράγματα, η πιθανή παραβίαση ευρεστεχνιών που καλύπτουν διάφορες πτυχές ε, φαρμακευτικών προϊόντων είναι ένα θέμα εμπορικό χωρίς επιπτώσεις για τον καταναλωτή. Στο ε, πρόταση κανονισμού λοιπόν θα έλεγα πως εμείς υποστηρίζουμε το προήμιο 17 για τα θέματα διέλευσης. Πιστεύουμε ωστόσο πως τα τελωνία χρειάζεται να έχουν κάποιες οδηγίες για να αξιολογήσουν τη δυνατότητα, την πιθανότητα μάλλον επιστροφής των αγαθών στην ευρωπαϊκή αγορά. Επίσης πιστεύουμε πως είναι σημαντικό ο αποστολέας και ο παραλήπτης των αγαθών να έχουν το δικαίωμα να ακουστούν και επίσης να ενημερωθούν για την κατάσχεση του προϊόντος τους ή για την παρακράτηση του προϊόντος τους. Όταν θεληφθεί δε τέτοιου είδους απόφαση είναι πολύ σημαντικό να ανακοινώνεται μέσα σε μια εργάσιμη ημέρα στον ε, αποστολέα και στον παραλήπτη, γιατί κάποιες φορές αυτό που συμβαίνει είναι ότι αγαθά σταματήσαν σε μια αποθήκη για δύο εβδομάδες και ο ιδιοκτήτης των αγαθών δεν το ξέρει καν γιατί κανείς δεν τον ενημέρωσε. Τέλος, πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό τα δείγματα να μην παίρνονται κατά τη διάρκεια της παρακράτησης. Είχαμε περιπτώσεις όπου λήφθησαν δείγματα, μετά υπήρξε κατάχρηση και ε, τα αποτελέσματα δεν είχαν καμία σχέση με τα παρακρατηθέντα αγαθά και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες ρήτρες ασφαλείας. Ε, τέλος, να σας πω επίσης ότι είναι σημαντικό και θα θέλαμε να ζητήσουμε τα φάρμακα να θεωρούνται αναλώσιμα αγαθά, ε, να μην τα κρατάνε πάνω από τρεις μέρες. Γιατί, γιατί ε, υπάρχουν πάρα πολλά αγαθά, τα οποία, ε, μάλλον φάρμακα, τα οποία είναι σημαντικό να μένουν στη σωστή αλυσίδα του κρύου. Αν δεν μπορούν να παρακατευθούν πάνω από πέντε μέρες, διαφορετικά είναι άχρηστα. Δηλαδή η καταπολέμηση της παραχάραξη, της παραποίησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εναντίον των θεμητών ε, φαρμάκων γενικευμένης ονομασίας. Ε, και δεν πρέπει αυτό να σχετίζεται με τι εγκληματικές ομάδες και τα εγκλήματα που διαπράττουν μέσω της παραποίηση ε, φαρμάκων θα πρέπει να κάνω έκκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην υπάρξει επιβάρυνση της πρόσβασης σε φάρμακα γενικευμένης ονομασίας. Σας ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα κάπως. Σας ευχαριστώ και εγώ. Είπατε πολλά σημαντικά πράγματα και οι διαφάνεια σας ήταν χρήσιμες. Τώρα, δίνω το λόγο στον Νίλ Νάριμαν αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Αθλητικών Ιδών και επίσης είναι παγκόσμιος διευθυντής πνευματικής ιδιοκτησίας της Πούμα. Ακούσαμε για τα προϊόντα πολυτελείας από τον Γερμανό συνάδελφο τώρα. Έχετε και εσείς να μας πείτε παρόμοια θέματα. Σας καλωσορίζω και σας δίνω το λόγο. Και εγώ σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλη τιμή κυρίες και κύριοι για μένα που βρίσκομαι εδώ, που έχω προσκληθεί να παρουσιάσω σε αυτή τη δημόσια ακρόαση το θέμα μας. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω γιατί για τον κλάδο μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετάσχουμε σε αυτή τη δημόσια ακρόαση με παρουσίαση. Η βιομηχανία αθλητικών ειδών ε, επηρεάζεται πάρα πολύ από τις απομιμήσεις, από το φαινόμενο το οποίο συζητάμε σήμερα, τις παραποιήσεις, απομιμήσεις, τα... τις μαϊμόδες. Είμαι εδώ εκ μέρους της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Αθλητικών Ειδών. Έχουμε 1.800 σήματα στην Ευρώπη. 11 ε, ομοσπονδίες εθνικές, βλέπετε εδώ ποιες, και συνολικά άμεσα ή έμεσα απασχολούμε πάνω από 640.000 Ευρωπαίους και κύκλο εργασιών έχουμε 65 δις. Το πολύ με την συνομοσπονδία μας μπορείτε εδώ να δείτε τα μέλη μας στις διαφάνειες. Θέλω όμως να σας μιλήσω για την πρόταση της Κομισιόν. Προτού ασχοληθούμε με το θέμα των προϊόντων σε διαμετακόμιση, transit δηλαδή, που είναι το θέμα αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να ασχοληθώ λίγο με την πρόταση της Κομισιόν στο σύνολό της. Πρώτα απ' όλα, είμαστε υπέρ της ευρείας κάλυψης των παραποιήσεων. Είμαστε υπέρ της κάλυψης του παράλληλου εμπορίου, πράγμα το οποίο δημιουργεί προβλήματα για τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και πρόβλημα ποιότητας στην ΕΟΧ. Ο βασικός λόγος όμως για τον οποίο υποστηρίζουμε αυτή την προσπάθεια της Κομισιόν είναι διότι ανακαλύπτουμε όλο και περισσότερα φορτία παραποιημένων αγαθών με, ανα... με με γνήσια. Είναι μια νέα συνήθεια αυτή, γνήσια με παραποιημένα αναμειγμένα. Τώρα, ως προς τη διαδικασία. Ε, η διαδικασία μας βοηθάει. Σήματα, βοηθάει σήματα σαν και τα δικά μας για να προστατεύσουμε τα πνευματικά μας δικαιώματα. Όμως υπάρχουν και ορισμένα σημεία τα οποία ανησυχούν πάρα πολύ τα μέλη μας. Θα σας πω ποια είναι. Το πρώτο σημείο είναι το εξής. Η πρόταση της Κομισιόν δεν δίνει καμία ευθύνη στους διαμεσολαβητές, όπως οι μεταφορείς, στους ενδιάμεσους δηλαδή. Είχαμε την παρουσίαση του κυρίου Βαν Μπέρ και είναι πολύ δύσκολο για μένα ε, να μην σχολιάσω τις απόψεις του. Ιδιαίτερα καθώς θεωρούμε ότι είναι πραγματικά άδικο να πέφτει όλο το βάρος του κόστους για την καταστροφή και την αποθήκευση στον ε, ε, ιδιοκτήτη του σήματος που δεν έχει καμία ανάμειξη στην παραποίηση. η ενδιάμεση όπως οι μεταφορείς, οι προωθητές κτλ. είναι πολύ πιο κοντά στους παραβάτες από ότι οι διοκτήτες σήματος. Οι δικαιούχοι δηλαδή. Και γι' αυτό δεν κατανοούμε γιατί δέχονται ότι γνωρίζουν τους αντισυμβαλόμενους αλλά δεν τους αποκαλύπτουν σε πολλές περιπτώσεις. Μπορώ να σας δώσω πολύ άριθμα παραδείγματα. Ακόμη και ο παραλήπτης ήταν ψευδής, ανύπαρκτος. Και δεν βάζουν κανένα όρο στις συμβάσεις τους, όπου, μέσω των οποίων να είναι υπεύθυνοι ο αποστολέας και ο παραλήπτης για όσα πραγματοποιούνται. Πραγματικά θα θέλαμε να υπάρχει μια διάταξη στον κανονισμό που τουλάχιστον να ρυθμίζει κάπως ε, ή να βάζει κάποιες ευθύνες και κόστη στους ενδιάμεσους. Τώρα, όσον αφορά το transit, είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό για την ε, βιομηχανία αθλητικών ειδών. Γενικά θα ήθελα να πω ότι εάν τα προϊόντα transit δεν σταματούν πλέον στα σύνορα της Ευρώπης μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα χρειαστεί να μιλήσουμε ε, για αυτό τον κανονισμό πλέον διότι θα υποφεληθούν οι παραποιητές ε, από αυτό το κενό στην νομοθεσία και θα στέλνουν τα πάντα transit. Μπορώ να σας δώσω πολλά παραδείγματα από άλλα μέρη του κόσμου. Νότια Αφρική, Μεξικό, οι παραποιητές χρησιμοποιούν αυτά τα κενά στο δίκαιο για να στέλνουν τα προϊόντα στους transit. Ε, ε, δεν θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση. αφόσον μιλάμε για απομιμήσεις, για λαθρεμπόριο ανθρώπων κτλ. Τι θέλω να πω τελικά. Ε, οι τελωνιακοί μπορεί να ανοίξουν ένα φορτίο και να βρουν μέσα λαθρομετανάστες για οι όπλα. Κανένας ε, δεν θα πει σε αυτή την περίπτωση όχι δεν μπορούμε να σταματήσουμε τα όπλα επειδή είναι τράνζιτ ή δεν μπορούμε να συλλάβουμε τους λαθρομετανάστες. Ε, λοιπόν, τι θα ήθελα. Θα ήθελα να αναθεωρήσετε τη σχετική διάταξη και να μας προστατεύσετε. Είναι σχεδόν αδύνατο για τους ε, δικαιούχους να αποδείξουν ε, ότι τα παραποιημένα πάνε στην ευρωπαϊκή αγορά το να δίνεται τη δυνατότητα να αποδείξει ο άλλος ότι είναι transit, αυτό μας δημιουργεί δυσχέρειες. Οι απαταιώνες επίσης, οι οποίοι εισάγουν προϊόντα, αν δεσμευτούν τα προϊόντα από τους τελωνιακούς, θα μπουν σε μία αποθήκη και θα απολυθούν τελικά σε μικρές ποσότητες χωρίς καμία εποπτεία από τους τελωνιακούς. Θα απολυθούν δηλαδή από την αποθήκη στην οποία θα δεσμευθούν. Θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Το 2008, 7% των συνολικών δεσμεύσεων ή κατασχέσεων τελωνία, από τα τελωνία ήταν transit εμπορεύματα. Το συνολικό ποσό απομιμήσεων ή παραπάνω, όχι με συγχωρείτε, διορθώνει ο μιλητής. 42% των παραποιημένων αγαθών βρέθηκαν στα 7% των δεσμευμένων φορτίων transit. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν δεν ελεγχόντουσαν αυτά τα φορτία transit, θα είχαμε χάσει την ευκαιρία να συλλάβουμε πάρα πολλά παραποιημένα. Τώρα, Όσον, αφορά τα δικαιώματα σήματος, ακούσαμε για τα φαρμακευτικά, για τα γενώσιμα φάρμακα και είναι πολύ σημαντικό να γίνει ένας διαχωρισμός στον κανονισμό μεταξύ γενικευμένης ονομασίας, ε, ευρεσιτεχνίας και σημάτων. Είναι διαφορετικά τα θέματα. Σύμφωνα με μία ρύθμιση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ινδίας και Βραζιλίας, συμφωνήθηκε να μην σταματά πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προϊόντα γενικευμένης ονομασίας. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με τα παραποιημένα. Είναι άλλο θέμα. Αυτά είχα να σας πω και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Well, thank you for, um, for some very clear and some very... Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σαφή παραδείγματα και σχόλια. Έχουμε καταλάβει κάπως καλύτερα την περιπλοκότητα του θέματος. Ο εισηγητής μας θα χρειαστεί να το σκεφτεί πολύ αυτό το θέμα που θίξατε. Λοιπόν, τώρα έχουμε και τους ειδικού μας. Ο κύριος Λουκ Ντεμπλίκ από, από την Ολλανδία, σύμβουλος τελωνίων, είναι στη ΜΕΑ της Ολλανδίας εδώ θέλουμε την άποψή σας από την πλευρά των τελωνιακών ορχών των κάτω χωρών. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να σας παρουσιάσω εδώ τα θέματα ε, πνευματικής συντεκτησίας σε ό,τι αφορά τα τελωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και πολύ επίκαιρο. Σας υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να κρατήσω το όριο ε, το χρονικό. Θα σας μιλήσω στα Ολλανδικά, αλλά οι συνάδελφοι στην Ολλανδία προτίμασαν και διαφάνειες στα Αγγλικά. Θα ξεκινήσω από το τέλος, με μία σύνοψη δηλαδή της παρουσίασής μου σε ό,τι αφορά πέντε σημεία. Πρώτον, δεδομένης, δεδομένων των συμφερόντων της ασφάλειας και της υγείας των καταναλωτών εκτός και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ολλανδία θεωρεί ότι θα πρέπει να διατυπωθεί ο κανονισμός ε, για την, ε, τα τελωνία. Δεύτερον, ε, στην αναδιατύπωση αυτή θα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητος ο ρόλος των τελωνίων. Τρίτον, η Ολλανδία συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η αναδιατύπωση θα πρέπει να περιλαμβάνει ε, το δικαίωμα των κατόχων και των ιδιοκτητών ε, των εμπορικών σημάτων. Κατά τέταρτον, η Ολλανδική νομοθεσία λαμβάνει υπόψη και των συμφέροντα τρίτων χωρών και πέμπτον θα πρέπει να, κατά την αδιατύπωση να δώσουμε σωστή ισορροπία μεταξύ μη φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων. Να σας εξηγήσω λοιπόν τι εννοώ. Θα ήθελα όμως να σας μιλήσω για τα τελωνία σε ό,τι αφορά τα πνευματικά δικαιώματα. Θεωρώ ότι είναι άσκηση ισορροπίας, ισοσκελισμού. Θα πρέπει να ισορροπήσουμε μεταξύ των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών των ε, δικαιωμάτων, πνευματικών δικαιωμάτων και των άλλων φορέων, όπως των μεταφορέων, για παράδειγμα. Αφενός, έχουμε μη εναρμονισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταξύ των κρατών μέλων και αφετέρου έχουμε εναρμονισμένους εκτελεστικούς κανόνες σε ό,τι αφορά τα τελωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρειάζεται να σας επισημάνω ότι μεγάλη πρόκληση κατά την ε, εφαρμογή του χαρακτήρα IPR αποτελεί και αυτό μια άσκηση ισορροπίας ε, στο διαδίκτυο. Ε, καταρχάς, τα τελωνία πρέπει να σκεφτούν θέματα υγείας και προστασίας του καταναλωτή και κατά δεύτερον, θέματα πνευματικής ιδιεκτοσίας του παραγωγού θα πρέπει τα θέματα αυτά να ενταχθούν ίσως και στο πλαίσιο των μικρών αποστολών, των μικρών δεμάτων. Προτού εστιαστούμε σε θέματα διαμετακόμισης, θα ήθελα να πω ότι δεδομένων των ε, διάφορων δύσκολων εγχειρημάτων που αναλαμβάνει το τελωνίο, ότι η αποτελεσματικότητα του ρόλου των τελωνίων σε ό,τι αφορά καταπολέμηση των ε, ε, παραβιάσεων ανθρωπινών δικαιωμάτων εξαρτάται από το κατά πόσο μπορεί να την δραματίζει ανεξάρτητο, αμερόληπτο ρόλο το τελωνίο. Θεωρώ ότι αυτό θα σημειωνόταν αν έπρεπε να αναλάβει νέες ευθύνες στα τελωνιακή αρχή. σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την επιβολή ενδεχομένων κυρώσεων. Τα μέτρα αυτά θεωρεί η Ολλανδία. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Ο ορισμός των παραποιημένων προϊόντων, όπως περιλαμβάνεται στην πρόταση. Ο ορισμός προβλέπει παραποιημένα προϊόντα είναι τα εμπορεύματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο ε, ε, εμπορίας και που παραβιάζει ε, μια εμπορική επωνυμία. Αλλά αυτό προϋποθέτει νομική δράση. Αυτό θα έφερνε την, τα τελωνία σε μια θέση που θα έπρεπε να αποφανθούν για το κατά πόσον υπάρχει παραβίαση και αυτό θεωρώ ότι δεν συνάδει με τον αμερόληπτο ρόλο που πρέπει να διδραματίζουν τα τελωνία. Συνολικά κρίνω, τον έφερε και ο εισηγητής ε, στα εισαγωγικά του σχόλια, θεωρώ ότι χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση για την αναδιατύπωση σε ό,τι αφορά την αλλαγή του ρόλου των τελωνίων. Αυτή η άσκηση ισορροπίας θεωρώ ότι είναι χρήσιμη και σε ό,τι αφορά τα προϊόντα σε διαμετακόμιση, γιατί η καταπολέμηση τέτοιων παραβιάσεων μέσω των τελωνίων σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει παρέμβαση στην ροή των προϊόντων και αυτό σημαίνει και προϋποθέτει δράσεις των τελωνίων, οι οποίες θα ήταν ασύμβατες με την ελευθερία διαμετακόμισης, όπως προβλέπεται στους διεθνείς εμπορικούς κανόνες από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μπορεί να σημαίνει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ αναπτυσσόμενων χωρών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με πρόσφατα παραδείγματα. Κάποια δέματα τα οποία κατήσχαν οι Ολλανδικές αρχές ε, σε ό,τι αφορά φαρμακευτικά προϊόντα αποτελούσαν παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Αλλά ίσως θα έπρεπε να αναζητηθεί μια νέα ισορροπία σε ό,τι αφορά τα πνευματικά δικαιώματα και το ρόλο των τελωνιακών αρχών. Θα σας ε, μιλήσω κι άλλο για το θέμα αυτό δεν θα σα μιλήσω για το παρελθόν, αλλά μόνο για το παρόν και το μέλλον. Αλλά θα ήθελα καταρχάς να τονίσω πόσο σημαντικό είναι και κάτι άλλο, μια, ένα άλλο στοιχείο για τα πνευματικά δικαιώματα. Η διατήρηση της σωστής συνεργασίας μεταξύ των κατόχων των δικαιωμάτων και των αρχών. Οι κανόνες θα πρέπει να διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο προκειμένου οι διοκτήτες των σημάτων να μπορούν να χρησιμοποιούν τα δικαιώματά τους, οπότε μπορούν να τα ασκούν. Και για να αποφευχθούν περιπτές καθυστερήσεις, να μην κάνουν τίποτα παραπάνω πέρα από αυτό. από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και στα τελωνία σημαντικές καθυστερήσεις και διαπιστώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της για να ακολουθεί αυτή τη διτή προσέγγιση στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2009 ξεκίνησε έναν διάλογο μεταξύ των θεσμικών των τελωνιακών αρχών και των εκπροσώπων της φαρμακοβιομηχανίας και κατάληξαν σε κοινέ δηλώσεις οι οποίες και καταγράφησαν στις κατοχώρες Η εκτέλεση από τις τελωνικές αρχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά διαμετεκόμιση επηρεάζεται ασφαλώς από την ομολογία σε ό,τι αφορά τα φάρμακα τα οποία κατασχέθηκαν το 2009. Αφενός ε, ε το δικαστήριο ότι δεν ε, μπορούσε να γίνει διαμετακόμιση, δεν μπορούσε να η διαμετακόμιση και μία πρόσφατη του ΔΕΚ, μιλάω για την υπόθεση Philips και Nokia, έριξε νέο φως ε, στην υπόθεση Ασφαλώς θα περιμένουμε την απόφαση τη δικαστική. Οι κατοχώρες θεωρούν ότι σε ό,τι αφορά τα νόμιμα γενώσιμα φάρμακα δεν είναι πιθανόν να καταλήξουν στην εσωτερική αγορά και ότι δεν τίθεται θέμα παραβίασης των ε, πνευματικών δικαιωμάτων και δεν θα έπρεπε να ευθύνεται το τελωνίο για τον έλεγχο αυτό. και σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε, να εξακολουθήσουμε να ακολουθούμε αυτή την πρακτική όσο του να υπάρξει καινούργια δικαστική απόφαση. Και αν υπομονούμε να ακούσουμε την ε, δικαστική απόφαση και το πώς θα δημορφωθεί μετά το ΡΙΚΑΣ, μετά από την αναδιατύπωση. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει περιθώριο συζήτηση σε ό,τι αφορά ε, προϊόντα τα οποία υποπτευόμαστε ότι αποτελούν παραποίηση από νομικής άποψης. Θεωρώ ότι πρέπει να διευκρινιστεί η θέση άλλων παραπημένων προϊόντων πέρα από τα φάρμακα και τίνω να συμφωνήσω με αυτά που είπε ο συνάδελφος από, το, από την Ίντα όταν είπε ότι πρέπει φαίνεται ότι ορίζονται διαφορετικά κριτήρια για διαφορετικές ομάδες προϊόντων στην αναδιατύπωση. Το θέμα είναι πώς θα βρούμε την ισορροπία μεταξύ της προστασίας των τρίτων χωρών σε ό,τι αφορά τα, τη διαμετακόμιση, γιατί αφενός ό,τι αφορά τα γενώσιμα φάρμακα έχουν συμφέρον να ε, δοθούν στην εμπορία τα ε, φάρμακα αυτά, αλλά αφετέρου όταν πρόκειται για παραποιημένα επικίνδυνα φάρμακα έχουν συμφέρον να εμποδιστούν. Δεν υπάρχει αρκετή σαφήνεια στην αναδιατύπωση, θεωρώ. Φυσικά είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε απόλυτα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου από αυτή την πλευρά να διαλευκανθεί η νομοθεσία και ακούσαμε και πολλές καλές ιδέες σήμερα. Ξεπέρασα κάπως τον χρόνο ομιλίας μου. Ελπίζω να μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή σύνοψη. Θα ήθελα εκ νέου να πω τα εξής, συνοψίζοντας πρώτον θέματα όπως η ασφάλεια και η υγεία των καταναλωτών εκτός και εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικά σε ό,τι αφορά την αναδιατύπωση. Δεύτερον, σε μια τέτοια αναδιατύπωση θέλουμε να διατηρηθεί ο μερόλεπτος ρόλος των τελωνιακών αρχών. Τρίτον, οι κατοχώρε συμφωνούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η αναδιατύπωση θα πρέπει, θα πρέπει να σημαίνει έναν ε, ε, ρόλο επαγρύπνησης για τον κάτοχο των ε, πνευματικών δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά τις, ε, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Θα πρέπει να βασιστούμε στην ομολογία και να λάβουμε υπόψη και τα συμφέροντα τρίτων χωρών. Και τέλος, κατά την αναδιατύπωση, θέλουμε να υπάρξει ισορροπία μεταξύ των εμπορικών σημάτων σε άλλες περιπτώσεις πέρα από τα γενώσιμα φάρμακα που βρίσκονται σε φάση διαμετακόμισης. Σας ευχαριστώ πολύ. Well, thank you very much for a very clear statement. Σας ευχαριστώ πολύ για τις αυτές σας δήλωση στο τέλος. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε αν όλοι οι αναλυτές τελικά συμφωνούν με τη σύνοψή σας, γιατί έτσι μας δίνεται κάποια βάση για να προχωρήσουμε. Με βάση περιπτώσει, ας δούμε αν έχουμε κάποια σύντομα ερωτήματα από του από τα μέλη. Όχι, έχετε κυρία Ρούλε κάτι να πείτε. Όχι. Ε, να κλείσουμε και αυτό το γύρο. Θα ήταν δίκαιο αν επαναρχόμουν στον κύριο Πούλεν αν έχει κάτι να πει για τις παρατηρήσει των άλλων και αν κάποιος άλλος θα ήθελε επίσης να το κάνει και μετά θα καλέσω την κυρία Ντερή να μας δώσει τη δική της παρατήρηση αντίδραση μάλλον στα όσα ακούσαμε για περίπου 5 λεπτά και μετά θα επανέλθω στον εισηγητή για να κλείσουμε την ώρα μας. Αν κάποιος άλλος ε, συμμετέχων θέλει να κάνει κάποιο σύντομο σχόλιο, ο κύριος Νιούμαν ζήτησε το λόγο. Α, ναι, θα έπρεπε να, ίσως να δώσω το λόγο και στην Πολωνική Προεδρία. Ο κύριος Σέντερς είναι εδώ. Και έχουν και άλλον ένα ομιλητή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. All right. Well, we'll see if we can fit you all in, if you all can be economical. Um, but let's just have a very brief reaction. Μια σύντομη αντίδραση από τον κύριο Πούλαν. Θα είναι ενδιαφέρον νομίζω αυτό, γιατί είχαμε ενδιαφέρουσε εισηγήσει. Θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε τι παρατηρήσει σα. Μάλλον πρέπει να μιλήσω μισό λεπτό. Τα όσα ακούσαμε νομίζω μας οδηγούν στο να κατανοήσουμε ότι υπάρχει συνένεση για το πώ πρέπει να προχωρήσουμε. Υπάρχει συμφωνία ότι υπάρχει σαφής ε, και υπάρχουν κίνδυνος από τα παραποιημένα προϊόντα, τόσο για τα προϊόντα διαμετακόμισης, όσο και για τα προϊόντα που κατευθύνονται στην ευρωπαϊκή αγορά και πρέπει αυτό να αντιμετωπιστεί. Επίσης, νομίζω προέκυψε το γεγονός ότι η νόμιμη ευρεσιτεχνία ή τα νόμιμα ε, ε, γενώσιμα αγαθά σε διακμετακόμιση θα πρέπει να μπορούν να προχωρήσουν και αυτό συμφωνεί και με τη δήλωση που έγινε από την EFPAA και από τον συνάδελφο των Ολλανδικών ε, Τελωνίων αναφέρθηκε αυτό, ότι συμφωνήθηκε και από τη φαρμακοβιομηχανία και από την ε, τις τελωνιακές αρχές. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι σαφές το τι πρέπει να κάνουμε εδώ. Εγώ θα ήθελα μόνο να προσθέσω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω τα τελωνία να έχουν τις σωστές ε, οδηγίες, κάποιες κατευθυντήριες γραμμές ή επικοινωνία μαζί μας για να έχουν ένα κατάλογο των ε, εταιριών που κατασκευάζουν τα φάρμακα αυτά δεν είναι και τόσες πολλές και αν έχουν κάποιο ύποπτο φορτίο να μπορούν να, μας, ε, να επικοινωνούν μαζί μας, να μην τα παρακρατούν άσχετα με το αν υπάρχει παραβίαση ευρεσιτεχνία ή όχι, ιδιαίτερα όταν είναι σε διαμετακόμιση. Και είναι πολύ σημαντικό οι τελωνιακέ αρχέ να στηριχτούν για να μπορούν πραγματικά να σταματήσουν τα πλαστά φάρμακα με ψεύτικο σήμα, παραχαραγμένο σήμα. Κύριος Νάριμαν, μια γενική παρατηρήση. Εγώ θα το εκτιμούσα αν τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου μέσω συζήτησης για την πρόταση έχουν υπόψη τους ότι η παραχάραξη είναι πραγματικά σοβαρό έγκλημα. Ο κ. Κριστόφ Ζήμερμαν ήδη μας μίλησε για τον αντίκτυπο στον καταναλωτή και του κινδύνου υγεία. Αυτό που δεν ανέφερε είναι πώς αυτά τα παραπημένα αγαθά κατασκευάζονται υπό ποιες συνθήκες περιβαλλοντικές, τι είδου συνθήκες εργασίας επικρατούν, παιδική εργασία εμπλέκεται εκεί, άνθρωποι που ασχολούνται με την καταπολέμηση της παραποίησης απειλούνται, δεν ανέφερε ότι η τελωνιακή υπάλληλοι που είναι υπεύθυνοι στο IPR για τα, δικαιω... τα πνευματικά δικαιώματα στο λιμάνι του Ντέρμπαν πυροβολήθηκε φέτος από Κινέζους ε, παραχαράκτες. Είναι σοβαρό έγκλημα. Δεν είναι κατανοητό για μένα και από την άποψη του καταναλωτή γιατί, να, γιατί πρέπει να συζητάμε για αγαθά παραποιημένα στις ε, βαλίτσες ε, των, ταξιδιωτών. Τα παραποιημένα αγαθά είναι παραποιημένα, είναι από μιμήσεις ούτως ή άλλως και πρέπει να δώσουμε μηνύματα στους καταναλωτές. Μιλάμε για εκστρατείες ενημέρωση των καταναλωτών γιατί θα ήταν λάθος μήνυμα αν για παράδειγμα δεν σταματάμε τα μικρά δέματα ή τα παραποιημένα αγαθά που περιέχουν οι βαλίτσες των ταξιδιωτών. Να επανέλθω στον κύριο Ντεμπέικα σε λίγο. Ο κύριος Νιούμαν θα πάρει πρώτο το λόγο και μετά ο κύριος Ντεμπλέικ. Κύριε Νιούμαν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Είχαμε την υπόθεση Nokia και η εταιρεία μου είχε ε, να υπερασπιστεί την Νόκια. Η υπόθεση δεν ήταν κάποιο εμπορικό κέρδος σε σχέση με την δέσμευση του φορτίου. Αυτό που αισθάνθηκε η Νόκια ήταν ελλείψεις της ρυθμίσης. Η απόφαση Νόκια θα καταλήξει την άλλη εβδομάδα, θα μας δοθεί μάλλον την άλλη εβδομάδα και έχουν αφαιρεθεί πολλά σημεία από τη νέα πρόταση. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ποια είναι η αντίδραση της Κομισιόν στον εισηγητή και γιατί τα προϊόντα transit ε, καλύπτονται από αυτή την πρόταση. Επίσης, Υπάρχει συνένεση μεταξύ όσων μιλήσαν σήμερα και θέλω, θα ήθελα δράση σήμερα ε, πάνω στο θέμα αυτό. Πρόεδρος. Τελευταίος ομιλητής ο κύριος Μπλέικ. Σας ευχαριστώ. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Να διαπιστώσω απλά ότι επικρατεί μεγάλη συνένεση για το ότι θα πρέπει να έχει τις σωστές αρμοδιότητες η τελωνιακή αρχή για να διαπιστώνει, για να μπορέσει να εκτελεί τα καθήκοντά της α, σεβόμενη τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων φορέων. Ευχαριστώ. Good. Well, I'm going Πρωτού δώσω τον λόγο στον εισηγητή, θα ήθελα τώρα να παρέμβει η Κομισιό και το Συμβούλιο, αν θέλουν. Ο κύριος Βελάσκο, αναπληρωτής τμήματάρχης, και η κυρία Καμάντρη από την DG Taxod και έχουμε και τον κύριο Σέντερ της Πολωνικής Προεδρίας. Παρακαλώ τα σχόλιά σας. Ας ξεκινήσουμε με τον κύριο Βελάσκο, Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Θα τελειώσουμε την Προεδρία. Κύριε Βελάσκο, ε, πέντε λεπτά μέγιστον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σχόλιο πολλών ομιλητών, την ανάγκη συνεργασίας με τρίτης χώρες και την ανάγκη ε, να πάμε στην πηγή. Αλλιώς συνεχώς τρέχουμε πίσω από το πρόβλημα χωρίς να το λύνουμε. Αυτή είναι μια δραστηριότητα ακριβώ τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Έχουμε εκτεταμένε δραστηριότητε, πρέπει να πω, στην προώθηση τη προστασία πνευματική ιδιοκτησία σε τρίτε χώρε, είτε πολυμερό στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, είτε πάλι μέσω διμερών διαπραγματεύσεων. Έχουμε διαπραγματευτεί συμφωνίες με πολλές χώρες και πάντα περιλαμβάνουμε κεφάλαιο πνευματικής ιδιοκτησίας προσπαθώντας να βελτιώσουμε την προστασία σε αυτές τις χώρες. Πολύ πρόσφατα το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει τη συμφωνία με την Κορέα. Τώρα έχουμε ε, τις συμφωνίες Περού, Κολομβίας και πολλών άλλων που θα φέρουμε μπροστά στο Κοινοβούλιο. Επίσης έχουμε ξεκινήσει διάλογο με τις προβληματικές χώρες. Είμαστε πολύ δραστήριοι στην Κίνα. Αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένα προβλήματα με τις τοπικές αρχές, φέρνουμε την βιομηχανία ε, να συμμετάσχει και πιέζουμε πολύ τα μέρη και η βιομηχανία μας ενημερώνει για τυχόν θετικά αποτελέσματα. Είναι δύσκολος ο αγώνας. Μιλάμε για τεχνικό και πολιτικό επίπεδο. Είναι συνεχής η διεργασία αυτή και δεν σταματάμε ποτέ. Τώρα, ο τελωνιακός κανονισμός θεωρείται υπόδειγμα ανά τον κόσμο. Είναι πολύ αποτελεσματικό εργαλείο, εμείς το υποστηρίζουμε στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και πολλές χώρες όταν θέλουν να βελτιώσουν το τελωνιακό του σύστημα το χρησιμοποιούν. Το προηγούμενο ήταν πολύ αποτελεσματικό μοντέλο. Τώρα θέλουμε το καινούριο να βελτιώσει πολλές πτυχές και να χρησιμοποιηθεί σαν πηγή έμπνευσης για την βελτίωση των προτύπων ανά τον κόσμο. Όσον αφορά το θέμα των προϊόντων γενικευμένης ονομασίας και των διαφόρων συμβάντων. Τα παρακολουθούμε πολύ κοντά για την Ινδία και τη Βραζιλία. Πάντα λέγαμε ότι ίσως ήταν σημαντικό να ρυθμίσουμε τον κανονισμό, αλλά δεν χρειαζόταν επανάσταση. Δεν κάναμε ποτέ κάτι εσφαλμένο, αλλά είμαστε σε επαφή για να φροντίσουμε το επεισόδιο να κλείσει μόλις εκδοθεί ο κανονισμός. Τελευταίο σχόλιο. Πάλι για την προώθηση της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες. Σύντομα το ε, Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει τη συμφωνία κατά της παραποίησης. Αυτό είναι ένα εργαλείο που θεσπίζουμε και να βελτιώσουμε την εφαρμογή της προστασίας σε τρίτες χώρες. Είναι σημαντικό μαζί με την εργασία για τον κανονισμό. Το Κοινοβούλιο πρέπει συνεπώς να θεωρήσει τη σύμβαση κατά της παραποίησης σαν ένα εργαλείο που κατατείνει στους ίδιους στόχους. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ακούσατε από την κυρία Χέντομπερτ ότι ήμασταν στη Σαντάη και όταν πήγαμε στην αντιπροσωπεία της Κομισιόν μας ενημερώσαν και πραγματικά πραγματοποιούνται πολλές προσπάθειες. Η κυρία Έντεριχ τώρα της Κομισιόν. Πέντε λεπτά maximum στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνήθως δεν μιλώ πολύ όπως γνωρίζετε. Σας ευχαριστώ που μας δώσατε την ευκαιρία να ακούσουμε όλα τα σχόλια που ακούσαμε σήμερα από τους ενδιαφερομένους για το θέμα των τελωνίων και της προστασίας των ε, πνευματικών δικαιωμάτων. Υπάρχει ευρεία υποστήριξη για την πρωτοβουλία της Κομισιόν και υπάρχει και αναγνώριση του ρόλου των τελωνίων στην προστασία. Νομίζω ότι η συζήτηση και οι παρουσιάσεις έδειξαν ότι διάφορες πτυχές που πρέπει να εξετάσουμε και όλα τα θέματα που προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτή την πρόταση είναι πολύ σχηδή. Ελπίζω ότι όλοι αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθήσαμε να βρούμε ισορροπία ανάμεσα στις διάφορες τοποθετήσεις των ενδιαφερομένων και λαμβάνοντας υπόψη και τα τελωνία. Μία ερώτηση μου έγινε συγκεκριμένη όσον αφορά τα μικρά φορτία ή δέματα. Θα ήθελα να σας πω ποια είναι η πρόθεση της Κομισιόν. Ο στόχος είναι να υποστηρίξουμε τα τηλωνία στις δυσκολίε που αντιμετωπίζουν λόγω της ποσότητας των μικρών δεμάτων που δεσμεύουν. Είναι ε, διαδικαστικό ε, το θέμα. Θέλω να καθησυχάσω τον κύριο Κορέα. Αυτή η πρόταση δεν σημαίνει ότι τα τελωνία θα ενεργούν μόνο σε περιπτώσεις μικρών φορτίων που θα οριστούν όποιο και αν είναι το μέγεθος των φορτίων τα τελωνία μπορούν να ενεργούν. Απλώς θέλουμε να βρούμε μια διαδικασία που να αντιμετωπίζει τα πολύ μικρά φορτία ή δέματα. Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης δείχνουν ότι είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να προσδιορίσουμε τι είναι ένα μικρό φορτίο ιδέμα. Όλοι ξέρουμε τι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά πρέπει να βρούμε τον ορισμό που θα λύνει το πρόβλημα και που θα διαρκέσει διαχρονικά. Προτείνουμε λοιπόν η Κομισιόν να έχει τη δυνατότητα να εξουσιοδοτήσει τον ορισμό για να συζητήσουμε με τους εμπειρογνώμονες. Έχουμε ήδη συζητήσει με τους εθνικούς εμπειρογνώμονες, αλλά δεν καταλήξαμε. 13 ιδέες μας δόθηκαν στην δημόσια διαβούλευση για τον ορισμό και δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε. Αυτό που είναι σημαντικό είναι αφήσουμε τη δυνατότητα να ενεργούμε γρήγορα σαν ανταπόκριση σε νέες τάσεις. Αν έχετε νέες τάσεις και ο ορισμός σας δεν σας βοηθά, τότε καθυστερούμε γιατί θα πρέπει να τροποποιηθεί και πάλι ο κανονισμός, πράγμα που σημαίνει χρόνο. Γι' αυτό με την εξουσιοδοτημένη πράξη πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να προσαρμοστούμε καλύτερα. Όσον αφορά την υγεία και τα φάρμακα, όπως είπε και ο κ. Στόλερ, πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ πολιτικής πνευματικής ιδιοκτησίας, υγείας και ασφάλειας των πολιτών. Και επισύρω το, την προσοχή σας ε, για την οδηγία, στην οδηγία ε, για τα παραποιημένα φάρμακα και που περιλαμβάνει μία διάταξη για τα transit. Έτσι θα μπορέσουμε να ενεργήσουμε για τα φάρμακα transit, τα οποία ε, είναι σημαντική υπόθεση. Όσον αφορά τη χρησιμοποίηση δεδομένων και πληροφοριών από εταιρείε και ε, τελωνία. Έχουμε το απόρριτο. Μην το ξεχνάτε. Αυτό είναι για την προστασία όλων των εταιριών. Αν θέλουμε να παρακλίνουμε από το απόρριτο, θα, θέλουμε να προσ... θα πρέπει να προσφύγουμε στην προστασία δεδομένων και τους σχετικούς κανόνες της ΕΕ και δεν νομίζω ότι είναι κάτι που θέλουμε σαν πολίτες της Ευρώπης. Αλλά αυτό δεν είναι στο χέρι μου. Όσον αφορά το transit, θα ήθελα να αποσαφηνίσω και πάλι ότι ακολουθήσαμε την ομολογία του δικαστηρίου. Τι μας λέει, έχουμε και τη γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα για την υπόθεση Νόκια. Το επίπεδο της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων εγγράφεται στον ουσιαστικό νομοθέτημα για το πνευματικό δίκαιο. Και εκεί πρέπει να δούμε ποιες είναι οι παραβολιάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι τελωνιακή νομοθεσία που δημιουργεί νέα δικαιώματα. Μπορούμε στον κανονισμό να πούμε μόνο ότι τα τελωνία μπορούν να ελέγξουν τα προϊόντα κάτω από όλες τις συνθήκες όταν είναι κάτω από την αποπτία τους. Όταν, όταν ασχολούνται με δέσμευση τότε θα πρέπει να αναφερθούν στο ουσιαστικό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ακούμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην Κομισιόν. Θυμόσατε ότι στην τελευταία ανακοίνωση για την εσωτερική αγορά είπαμε ότι θα αποσαφηνίσουμε το θέμα των προϊόντων transit. Και αυτό είναι το έργο των συναδέλφων μου στη Γενική Διεύθυνση Αγοράς τώρα. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Θα αναφερθούμε σε κάποια άλλα ζητήματα τα οποία ε, ασφαλώς και ε, απασχολούν ιδιαίτερα τον εισηγητή. Και χαίρομαι που έχουμε μαζί μας και την πλονική προεδρία. Θα σας δώσω το λόγο για καταληκτικά σχόλια. E, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Θα ήθελα λοιπόν να σας μιλήσω για τις δικές μας δραστηριότητες. Να αναφερθώ και σε κάποια θέματα τα οποία ακούσαμε. Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να συμμετάσχω στην ε, δημόσια ακρόαση αυτή. Πολλές ε, σημαντικές παρουσιάσεις έγιναν. Ακούσαμε και πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, πολλέ ενδιαφέρουσε πληροφορίε. και σίγουρα θα χρειαστεί να τα επεξεργαστούμε στο Συμβούλιο σε ό,τι αφορά και το έργο μας για τον κανονισμό για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Πολλά θέματα θα πρέπει να εξεταστούν εντελεχώς. Πολλά θέματα τα οποία έχουν ήδη συζητηθεί και όπως και εσείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμείς στο Συμβούλιο εξετάζουμε όλες αυτές τις πτυχές ακολουθώντας συχνά παρόμοιες προσεγγίσεις και εντοπίζοντας παρόμοια προβλήματα όπως μας ανέφερε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα μικρά δέματα, το πρόβλημα των ορισμών όπως μας ανέφεραν και οι εμπειρογνώμονες είτε μέσω κανονισμού είτε μέσω πράξης κατεξουσιοδότησης και εμείς έχουμε κάνει τέτοιες σκέψεις και βάσει της διαδικασίας συναπόφασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξουμε σε ένα τελικό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά και το θέμα των ε, αποσκευών των ταξιδιωτών. Θα πρέπει να μεταχειριζόμαστε, πώς θα πρέπει να μεταχειριζόμαστε τις αποσκευές και τα προϊόντα απομίμησης που βρίσκονται σε αυτές τις αποσκευές. Θα πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή, θα πρέπει να προχωρούμε σε κατάσχεση όλων των προϊόντων. Είναι δυνατόν να γίνει αυτό ή θα πρέπει να είμαστε πιο ελαστικοί. Γεννάται και το θέμα του κόστους καταστροφής των μικρών αυτών δεμάτων. Ποιος ε, πρέπει να φέρει την ευθύνη για το κόστος αυτό. Πολλές και διαφορετικές είναι οι απόψεις. Άλλοι λένε ότι οι τελωνιακές αρχές δεν είναι έτοιμες στην παρούσα φάση για να αναλάβουν το κόστος αυτό. Επίσης και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Στην παρούσα φάση στο Συμβούλιο έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει το πρώτο σχέδιο κειμένου για τον κανονισμό για την ανταγωνιστικότητα στις 5 Δεκεμβρίου. Θα συζητήσουμε την έκθεση προόδου που έχει προετοιμάσει η Πολωνική Προεδρία και ελπίζω ότι το Δεκέμβριο θα ξεκινήσει η πιο στενή συνεργασία με τους εισηγητές και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου γρήγορα να προχωρήσουμε κατά τη διάρκεια της Πολωνικής και της Δανικής Προεδρίας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ νέου για την ευκαιρία που μου δώσατε να ακούσω όλα αυτά τα ενδιαφέροντα σχόλια, όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Ασφαλώς και θα τα λάβουμε υπόψη κατά την κατάρτιση του κοινού κανονισμού για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων σε σχέση με την εφαρμογή του από τις ελληνικές αρχές. Ευχαριστώ, ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Χαρήκαμε που είσαστε κι εσείς εδώ όλο το απόγευμα. Σας εύχομαι καλά αποτελέσματα και ο κύριος Κρόιτσμαν και σε επαφές με τον κύριο Κρόιτσμαν. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε κύριε Κρόιτσμαν για τη διοργάνωση της ακρόασης. Κάντε παρακαλώ κάποια καταληκτικά σχόλια. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ Μάλκολμ αποδείχτηκε ότι η ακρόαση ήταν πάρα πολύ σημαντική και ήταν σωστό το ότι διοργανώθηκε. Τρία σημεία θα ήθελα να αναφέρω συνοπτικά. Αυτά που μας είπε ο Γερμανός Αντιπρόσωπος για το πώς θα πρέπει η διαδικασία μεταξύ των δικαιούχων και των καταναλωτών να βελτιωθεί. Δεύτερο σημείο, νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε το πρόβλημα ορισμού του μικρού δέματος. Λάβουμε προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξουμε σε έναν κοινό ορισμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει κάθε παραποιημένο προϊόν να διώκεται. Το ίδιο ισχύει και για τις αποσκευές οι οποίες στην παρούσα φάση δεν συμπεριλαμβάνονται. Δεν έχει νόημα να ορίσουμε τα μικρά δέματα και να πούμε ότι αυτά επιτρέπονται. και να επιτρέπεται να μεταφέρει ο επιβάτης οτιδήποτε πάνω του στις αποσκευές του. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ρυθμιστεί αυτό. Επίσης κάτι άλλο που είναι πολύ σαφές, το θέμα των εμπορευμάτων σε διαμετακόμιση. Θα πρέπει να επιληθεί. Δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουμε Όπω είπε και η σε ό,τι αφορά τα γενώσιμα, κατά τα άλλα θα πρέπει να διώκονται. Δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης των γενώσιμων. Ο συνάδελφο από το Ολλανδικό ε, Υπουργείο ανέφερε ότι αυτό είναι απόλυτα δυνατόν. Αυτά νομίζω ότι θα αποτελέσουν μια πολύ καλή βελτίωση της πρότασης κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος. Για να κλείσω, να σας πω ποιο είναι το χρονοδιόγραμμά μας σε ό,τι αφορά το Κοινοβούλιο. Ο εισηγητής ασφαλώς και θα λάβει υπόψη όλο το υλικό το οποίο ακούσαμε σήμερα. Θα μας αποστείλει τις προτάσεις του 8 Δεκεμβρίου για μετάφραση. Θα τη συζητήσουμε μετά το Χριστούγεννα, τον Ιανουάριο. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 19η Ιανουαρίου και είμαι βέβαια ότι θα δραστηριοποιηθείτε όλοι σας. Θα εξετάσουμε 6 Φεβρουαρίου τις τροπολογίες και προγραμματίζεται η ψηφοφορία στην Επιτροπή στις 28 Φεβρουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε έτοιμοι για ψηφοφορία στην Ολομέλεια 28-29 Μαρτίου. Ανάλογα και με τις ε, εξελίξεις στο Συμβούλιο σε περίπτωση που θέλει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις η Δανέσικη Προεδρία. Αυτό όμως από πλευράς του εισηγητή. Ήταν νομίζω πολύ καρποφόρο το απόγευμα και η ακρόαση να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες για το υλικό, το πολύ πολύτιμο που μας παρουσίασαν και ελπίζω να παραμείνετε σε επαφή μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Προφανώς και θα συνεργαστούμε και με τους σκιώδες και με τις πολιτικές ομάδες και με τις δύο άλλες συναρμόδιες επιτροπές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους ακροατές στο διαδίκτυο γιατί υποπτεύουμε ότι πολλοί θα παρακολούθησαν αυτή την ακρόαση. Internal Market Committee website and signing up for that. We're always very pleased to have new readers. Και επίσης τα λάβατε και το ε, ενημερωτικό δελτίο μας ε, στο διαδίκτυο που θα σας ενημερώσει και για τις μελλοντικές μας συνεδριάσεις οι οποίες επίσης αναμεταδίδονται ηλεκτρονικά. Σας αφούμε λοιπόν καλό απόγευμα και σας ευχαριστώ πολύ. Oh, and thank you very much to our hard-working interpreters as always.